Okay, colleagues, can I... Συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Can I, um, start with the report by... Θα ξεκινήσω ενημερώνοντάς σας για τη συνεδρίαση των συντονιστών και τις ανακοινώσεις του Προέδρου. Okay, Καθορισμένος, καθορισμός των εισηγητών και των συντακτών κειμένων. Είχαμε μια έκθεση όσον αφορά τον κανονισμό που τροποποιεί τον, 100, 1406 που δημιουργεί την υπηρεσία θαλασ... ασφαλείας θαλασσίων μεταφορών. Οι συντονιστές αποφάσισαν η ομάδα S&D να καθορίσει τον εισηγητή. Όσον αφορά τη γνωμοδότηση που τροποποιεί την οδηγία 25 του 2000 όσον αφορά τις διατάξεις για ελκυστήρες που διατίθενται στην αγορά σύμφωνα με το σχήμα, με το πλαίσιο ευελιξίας. Στον Στονιστέρα αποφασίσαν κύριε να αναλάβει αυτή την γνωμοδότηση. Ως και η τροποποιούσα οδηγία ακολουθεί την ε, ίδια προσέγγιση για τις ακίνητους, ε, ακίνητα μηχανήματα, σταθερά μηχανήματα για τους δρόμους Και προσθέτουμε λοιπόν και αυτή την γνωμοδότηση σχετικά με τους ελκυστήρες, τρακτέρ. Άλλα έγγραφα που ελήφθησαν, προς, παρελήφθησαν και εξετάσαν συντανιστός, η έκθεση για την θαγένεια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως 2010 που αφαιρεί τα εμπόδια για τα δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Οι συντονιστές αποφάσισαν να μην γίνει τίποτα Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς ενιαία αγορά, πράξη ενιαία αγοράς για πολύ ανταγωνιστική ε, και οικονομία και κοινωνική οικονομία. Λάβαμε επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής ΕΜΚΟ, του κ. Μάλκομ Χάρμπορ. Κάλεσε την Επιτροπή μα να υποβάλει νομοδότηση επί νομοθετικών προτάσεων βάσει των αποκλειστικών νομοδιοτήτων μα. Συμφώνησα, συντονιστέ με την πρόταση του Προέδρου να υποβάλουμε γνωμοδότηση υπό τη μορφή επιστολής, δική μου, απευθυνόμενη προς τον κύριο Χάρμπορ, συμπεριλαμβάνωσα σχόλια ενδεχομένως των συντονιστών. Και αυτή η διαδικασία είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να περάσουμε μια γνωμοδότηση στην ΙΜΚΟ καιρό. σύμφωνα το χρονοδιάγραμμα, διότι η ΙΜΚΟ προέβλεπε ότι θα ολοκληρωθεί το θέμα μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Οπότε προτάθηκε ο πρόεδρος να στείλει επιστολή υπομορφή γνωμοτήσεω προς τον πρόεδρο τη Επιτροπή και η επόμενη συνεδρίαση συντονιστών θα συζητήσει την επιστολή και θα συμφωνηθεί και ένα κοινό κείμενο. Τώρα σε ανακοίνωση για ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική για την εποχή τη παγκοσμιοποίηση, δεν ελήφθη απόφαση και το ίδιο για τις ε, άλλες δράσεις μέχρι την ε, αριθμό 11, προπολογισμό του 2012, απόφαση των συντονιστών ήταν η ομάδα S&D να καθορίσει τον εισηγητή για την ε, διαδικασία του προπολογισμού του 2012. Είναι η κυκλική εναλλαγή. εναλλαγή. Ο κύριος Ρίκε είναι εισηγητή για τον προπολογισμό 2011. Θα συνεχίσει το έργο του για τις υπόλοιπες φάσεις λόγω διαδικασίας μέχρι ότου να επιληθούν. Ντόμινι Ρίκε θα συνεχίσει με τον προπολογισμό 2011 μέχρι να ολοκληρωθεί αυτό και μετά τον προπολογισμό του 2012 τον αλάβει η ομάδα S&D που θα καθορίσει η συγγητή. Όσον αφορά το μέλλον το, της χρηματοδότησης του 10T αποφάσισε οι συντονιστές να καλέσουν τη Γενική Διεύθυνση την Αρμόδια και τους διάφορους φορείς να συζητήσουν τη μελλοντική την ε, χρηματοδότηση τον λόγο προγράμματο και να προετοιμαστεί και ένα έγγραφο εργασίας υπό την ευθύνη του Προέδρου που θα συζητηθεί στην Επιτροπή και με τη συνδρομή των άλλων αρμοδίων επιτροπών. Σε αφορά την επιτροπολογία, η Αντιπρόεδρο Τικάου αναφέρθηκε στο πρόγραμμα εργασιών για το 2011. Θα, η συνέχεια θα εξαρτηθεί από τις περαιτέρω της Επιτροπής Ήτρε. Στα διάφορα οι συντονιστέ είχαν στο φάκελό του την ανταλλαγή επιστολών μεταξύ τη Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και τη Επιτροπή Μεταφορών, του Προέδρου τη Επιτροπή Μεταφορών, σχετικά με το αίτημα τη Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών να συμμετάσχει στην έκθεση ιδίας πρωτοβουλία του κυρίου Ντεγκράνδε Πασχουάλ όσον αφορά την ασφάλεια των αερομεταφορών σύμφωνα με τη διάταξη 51, με το άρθρο 51. Η πρόταση θα διαβαστεί στη διάσκεψη των Προέδρων προ λήψη αποφάσεω, γιατί όπω γνωρίζετε έχουμε κάθετα αντίρρηση στο η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών να μπει βάσει του άρθρου 51 να παρισφρήσει τις εργασίες μας. Θα αποφασίσουν τώρα οι πρόεδροι στη διάσκεψη των πρόεδρων των Επιτροπών. Η συνάντηση με τα παλιά μέλη της Επιτροπής Μεταφορών να σας υπενθυμίσω ότι θα υπάρξει ε, με τη συνάντηση με την Κεντρική Επιτροπή για το Ρήνο την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου στο Στασβούργο από τις 2 μέχρι τις 4 ε, θα επισκεφθούμε την Επιτροπή για το Ρήνο. Όλα τα μέλη που ενδιαφέρονται για να πάνε στη συγκεκριμένη επίσκεψη, παρακαλώ γνωστοποιήστε το στην γραμματεία, ούτως ώστε να γνωρίζει και η Επιτροπή για το Ρήνο πόσοι θα καταθάσουν. Θα υπάρξει έκτακτη συνεδρία Επιτροπής Μεταφορών τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου από τις 7 μέχρι τις 8.30 στο Στρασβούργο. Ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Κάποιοι από εσά ίσως να προσπαθείτε να αποφεύγετε απελπισμένα τη συνεδρία των Επιτροπών μας στο Στασβούργο, τη Επιτροπή μα στο Στασβούργο. Πρέπει να πραγματοποιηθεί, θα συμμετάσχει ο Πρόεδρος Κάλλας, ο οποίος θέλει διακαώς να μας μιλήσει τα αποτελέσματα του άτυπου συμβουλίου που θα συζητήσει το TNT στη Βουδαπέστη το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. η κυρία Τσικάου, η αντιπρόδοση κυρία Τσικάου, εκπροσώπησε την Επιτροπή Μεταφορών στην ΣΤΟΑ, στο πάνελ ΣΤΟΑΣ και ενημέρωσε του συντονιστέ για την ετήσια έσκεψη ΣΤΟΑ για εκοκινητικότητα στι 7 Δεκεμβρίου που θα γίνει. Όσον αφορά την Ευρωβινιέτα, ο εισηγητή, ο κ. Αλκαντράου, ενημέρωσε του συντονιστέ όσον αφορά τι ερευνητικέ συνομιλίε του με τη Βελγική Προεδρία. Η θέση του Συμβουλίου θα διαβιβαστεί στο Κοινοβούλιο μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου και ο εισηγητής θα συναντηθεί με τους σκιώδεις εισηγητές της 7 Δεκεμβρίου για να καθοριστούν τα βασικά σημεία για τις άτυπες διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο που θα ξεκινήσουν τον ε, Ιανουάριο του επομένου έτους και μετά θα μας ενημερώσει θα ενημερώσει την πλήρη επιτροπή τον μήνα Ιανουάριο και οι συντονιστές ε, ενέκριναν την έκθεσή του και την ε, λόγο προσέγγιση. Αυτά όσον αφορά τις συνεδρίες των συντονιστών και τις ανακοινώσεις του Προέδρου. Υπάρχει κάποιος που έχει ερωτήσεις, κάποιο σημείο που θέλει να θίξει. Εάν δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, μπορούμε λοιπόν να συμφωνήσουμε όσον αφορά τα όσα υπόθηκαν και ότι ενημερωθήκατε. Μετά πάμε στις ψηφοφορίες. Έχετε όλοι τους κατα... τις κάρτες σας των ψηφοφοριών. Να κάνουμε ένα ανέλεγχο, μια δοκιμή. Έτοιμοι για τη δοκιμή. Ξεκινάμε λοιπόν τη δοκιμή, δοκιμαστική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Εντάξει, άναψε. Δεν είναι προσωπικό, Μάικλ. Απλώς το, το κόψαμε το μηχάνημά σου στο βράδυ. Το κλείσαμε. Δουλεύει τώρα, Μάικλ. Ωραία. Ψηφίσατε όλοι. Μισό λεπτάκι. στις υφοφορίες. Όλα εντάξει. Κυρία Κάστανιτς, δεν έχουμε παραπάνω μέλη για κάποια ομάδα που ψηφίσουν. Έχουμε και έναν βουλευτή, τον κύριο Σασόλη, ο οποίος δεν έχει ακόμα την κάρτα του, εντάξει. Ξεκινάμε με την έκθεση ΚΟΡΚ, Συμφωνία Υπηρεσιών μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Δικαιοδεφυγική Οικονομική Νομισματική Ένωση σχετικά με ορισμένε στεγέ των αεροπορικών υπηρεσιών. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 32 ψήφισαν, 32 υπέρ. Χωρίς αποχές και χωρίς αρνητικές ψήφους. και 33 με την μία που λείπει. Κυρία έκθεση Ρόσμπαχ. Νομίζω ξίσου εύκολα θα προχωρήσει όπως και οι προηγούμενη. Α, όχι. Ωραία πρόγραμμα για το Ευρωπαϊκό Αστικό Περιβάλλον μέλο στο πλαίσιο τη πολιτική συνοχή. Η κυρία Ρόσμπαχ είναι η συγγήτρια. Ξεκινά με τροπολογία 7 που υπευλήθη από τον κύριο Ζέλερ υπέρ. Κατά αποχέ. εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Σαν προσθήκη προφορική τροπολογία τη εισηγήτρια. Να μπει σαν νέα σε αυτή η προσθήκη. 1α. Υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά σε ελέγξουμε. Να πάρω και μια ιδέα ποιε είναι οι ισορροπίε. Τροπολογία, έξι προφορική τροπολογία σαν προσθήκη. Ξεκινάμε την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Τέλος. Δεκαπέντε υπέρ, 19 κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 9, σαν λόβα σαν προσθήκη Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά θα κάνουμε έλεγχο. Τροπολογία 9, ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, τέλος ψηφοφορίας. Δεν θα κάνει διαφορά. 20-14 θα ήταν, έτσι κι αλλιώς περνάει, εγκρίνεται. Ο κ. Κάντσεν ακόμα διαπραγματεύεται, το έμεινε από χθε το βράδυ, συμβιβαστική Β. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, άρα η 8 κατά πίπτη. 10. Κατά τμήματα, δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα μέχρι αρχή της επικουρικότητας. Δεύτερο τμήμα από το τονίζει. Λοιπόν, για το πρώτο τμήμα μέχρι την αρχή της επικουρικότητας υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές και αυτό εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 12 κατέπεσε, 13 κατά τμήματα, πρώτο τμήμα μέχρι εμπλεκόμενοι, stakeholders υπέρ του πρώτου τμήματος και που λέει stakeholders, διαφερόμενοι, εμπλεκόμενοι, κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα λαμβάνοντας υπόψη και λοιπά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική C λατινικό υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 22. Οι άλλες καταπίπτουν κατά τμήματα αποδείχνει μέχρι πιο ευάλωτη χρήση των δρόμων. Δεύτερο τμήμα μετά, αυτό που ακολουθεί. Λοιπόν, το δεύτερο τμήμα θα καταπέσει αν το πρώτο τμήμα καταπέσει. Απορριφθεί μάλλον. Λοιπόν, πρώτο τμήμα υπέρ. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πρώτο τμήμα υπέρ. Υπέρ του πρώτου τμήματος κατά αποχές εγκρίνεται. Άρα πάμε στο δεύτερο, το υπόλοιπο υπέρ κατά έλεγχος για το δεύτερο τμήμα. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Δεκαεπτά με 17 δεν εγκρίνεται. Συμβιβαστική D λατινικό υπέρ. Α, συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. 23, ζητώ συγγνώμη. 23, πρώτο τμήμα. Σε επίπεδο αστικό, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα. Παρατρίνιο που ενδείκνεται υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική D λατινίκο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 29. Αυτή η τροπολογία εν μέρη καλύπτεται από τη συμβαστική D, αλλά θα πρέπει να ψηφίσουμε. Σαν προσθήκη, βάδισμα, ποδηλασία, δημόσιες μεταφορές, μοίρασμα αυτοκινήτου, κοινή χρήση αυτοκινήτου, υπέρ, κατά, αποχές, ας ελέγξουμε. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. 16 υπέρ, 18 κατά, απορρίπτεται. 25 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 30 βαντάλεν υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 31, 31 για Λεσέντερ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά αποχές ας γίνει έλεγχος για την 35 ξεκινάμε η ευτής είναι μπορείτε λοιπόν από την ομάδα αυτή να αφαιρέσετε μια κάρτα έχετε έναν παραπάνω έχετε μόνο μία ψήφο. Αν βγάλετε τη δική σας κάρτα, πω μαγεία. Τέλος ψηφοφορίας. 14 υπέρ, 19 κατά, απορρίπτεται, 36 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 37 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 38, τέσσερα τμήματα. Πρώτο τμήμα, μέχρι βιώσιμο. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, η κατανομή των πόρων της συνοχής για τους ιδιοδρόμους και υπέρ, κατά, αποχές Απορρίπτεται. Μάικλ, συζήτησε με τελείωσε ψηφοφορίε. Απορρίπτεται, λέω. Γράψε εξήγηση ψήφου μετά. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τέταρτο τμήμα. 15% για προγράμματα για βάδισμα κλπ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 39. Ρόσπαχ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 40 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 42 σε δύο τμήματα όλο το κείμενο εκτός από τη φράση εξετάζοντας τη δυνατότητα να διευρυθεί το πεδίο εφαρμογής των δικαιωμάτων αστικής κινητικότητας. Πρώτο τμήμα χωρίς αυτές τις λέξεις υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα το υπόλοιπο υπέρ κατά αποχές έλεγχος για το δεύτερο τμήμα σας παρακαλώ ξεκινάμε ψηφίσατε όλοι τέλος 15 υπέρ, 19 κατά, απορρίπτεται 44 υπέρ, κατά, αποχές, Έλεγχος για τη 44. Ξεκινάμε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Εγκρίνεται 17 υπέρ, 16 κατά. 43 Τσικάου υπέρ, κατά, αποχές. Ξανά και εδώ έλεγχος για τη 43 σαν προσθήκη. Ξεκινάμε. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Εγκρίνεται 18-16-45. Καταπίπτει. 46 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 47 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 55 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. Πάμε σε τελογικές σκέψεις. Συμβαστική α. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 1, η 3, η 2 καταπίπτουν. Συνεπώς 4 τώρα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται πέντε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Ξεκινάμε. Μισό λεπτό. υπομονή. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Τέλος. 33 ψήφισαν, 32 υπέρ, μία ψήφος κατά. Κανονικά είναι 33 υπέρ, μία ψήφος κατά. Εγκρίνεται συγχαρητήρια κυρία Ροσμπαχ. Well done, Okay, we go on to the next item on the agenda. Mr. Zasa... Πάμε στο επόμενο σημείο της ημέρης της διάταξης. It gives you five minutes to... Πέντε λεπτά θα σας δώσω για να αποχωρήσετε ησύχως. Κύριε Λάιτφριντ, ε, θέλετε να πείτε κάτι? Όχι. Βαζεσάρε, okay. So we'll just wait. We're minutes ahead of time because you... Επειδή ήμασταν τόσο αποδοτικοί, έχουμε γλιτώσει και πέντε λεπτά. Οπότε, σας δίνω πέντε λεπτά να ξεκουραστείτε. Ο κύριος Κάντζεν και εγώ θα πάμε να διαπραγματευτούμε έξω και θα τα ξαναπούμε σε πέντε λεπτά. Okay, colleagues. transport agreement between... Συμφωνία αεροπορικών μεταφορών, αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ΕΠΑ. Ο κύριος, Ζασα... ο κύριος Ζασάντα είναι ο εισηγητής. Η, η Ολομέλεια ενέκρινε όμως στις 17 Ιουνίου ένα ψήφισμα για, τις, ε, για τους περιορισμούς των επενδύσεων και ζητά να συνεχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Για να το έχετε υπόψη σας, σας το λέω. Ο κύριος Ζασάντα είναι ο εισηγητής μας. Πού είναι? Που... Α... Κύριε Ζασάντα, έχετε το λόγο. Dziękuję bardzo za głos. Chciałbym, aby Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ακούσω και τις δικές σας ε, απόψεις για τη δεύτερη φάση της συμφωνίας των αεροπορικών μεταφορών μεταξύ Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης και ΕΠΑ. Η συμφωνία αυτή όντως είναι πολύ σημαντική γιατί οι αεροπορικές αγορές και των δύο χωρών συμβάλλουν κατά 60% στο, στην παγκόσμια αγορά. Εμείς είμαστε θύμα της διαδικασίας, γιατί η σιωπηρή διαδικασία δεν μας έδωσε την ε, νομική ε, ισχύ που θέλαμε, οπότε εμείς απλώς ένα ναι ή ένα όχι μπορούμε να πούμε ως κοινοβούλιο. Να σας πω κάποια στοιχεία η βασική συμφωνία εφαρμόζεται από το 2002 και περιλαμβάνει μια ρήτρα σύμφωνα με την οποία εάν δεν ξεκινήσει η δεύτερη φάση μέχρι το Νοέμβρη του 2010 τότε ακυρώνεται η συμφωνία. Παρ' όλα αυτά το πρωτόκολλο έχει υπογραφεί αλλά δεν εφαρμόζεται. Η αρχική συμφωνία και εδώ θα ήθελα να σα ευστήσω την προσοχή σε μια πολύ καλή ε, έκθεση ενό συναδέλφου. Αυτή η συμφωνία ήταν το πρώτο βήμα για μια ενισχυμένη συνεργασία που ήταν δεσμευτική και για τα δύο μέρη, για διάφορου τομεί, απελευθέρωση, επιπλέον δυνατότητες επένδυση, περιβαλλοντική προστασία, υποδομέ. Ε, αεροπορικές. Ευρεία ε, πρόσβαση σε εναέριες μεταφορές και διαθεσιμότητα των αεροσκαφών με πλήρωμα. Σας προτείνω λοιπόν τώρα να επικεντρωθούμε σε κάποια βασικά σημεία. Ο τελικό στόχος της συμφωνίας είναι η απελευθέρωση τη αγορά. Οπότε τίθεται το ερώτημα η συμφωνία έτσι όπως έχει εκπονηθεί ε, μας βοηθά να επιτύχουμε το στόχο μας. Επίσης, έχει γίνει υπερκής πρόοδος ό,τι αφορά τον, την άρση των περιορισμών που υπάρχουν στην αμοιβαία συμφωνία, άρθρο 21 ας πούμε. Και τρίτον, το πρόγραμμα Fly America είναι καλή απάντηση στα όσα έχουν θέσει ως προβλήματα οι Αμερικανοί, άρθρο 7 για παράδειγμα. Η συμφωνία αυτή καθ' αυτή είναι καλή και για τις δύο πλευρές. Θα πρέπει βεβαίως να ε, ξεκινήσουμε και την τρίτη φάση των διαπραγματεύσεων. Αυτά πρόεδρε από μένα και ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Πριν δώσουμε το λόγο στα, στους συναδέλφους, ε, να ακούσουμε τον κύριο Καγιάκα και μετά να ακούσουμε και, τον, ε, και τους υπόλοιπους, να ακούσουμε πρώτα την Κομισιόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Ζασάντα για τα σχόλιά του και τα μέλη της Επιτροπής σας για την βοήθεια που μας δώσατε για αυτή τη δύσκολη διαπραγμάτευση με, τους, με τη ΣΥΠΑ για τις εναέριες μεταφορές. Οι διαπραγματεύσεις αυτές έχουν γίνει τα τελευταία 7 χρόνια σε 19 γύρους. Η συμφωνία που συζητάτε σήμερα είναι η δεύτερη φάση ήταν ε, ενεκρίθη ομόφωνα από όλους τους Υπουργούς Μεταφορών στις 24 Ιουνίου και πρέπει να πω ότι και οι δύο πλευρές ε, του Ατλαντικού έχουν δώσει πολύ θετικά σχόλια ε, και, τα, και οι αεροπορικοί σταθμοί και οι ενδιαφερόμενοι φορείς και οι αεροπορικές εταιρείες που συμμετείχαν ενεργά σε όλες αυτές τις διαπραγματεύσεις. Τι είναι σημαντικό τώρα για αυτή τη συμφωνία είναι ότι συνεχίζει τη διαδικασία συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΠΑ. Και το κάνει με μια προσέγγιση αγορά προς αγορά. Δεν μιλούμε δηλαδή για 27 μεμονωμένες χώρες με διμερείς σχέσεις, μιλούμε για μία ενιαία σχέση η οποία συνδέει την ευρωπαϊκή αγορά με την αμερικανική. Και όπως είπε ο κύριος Ζασάντα, έχει απελευθερώσει το 60% των παγκόσμιων μεταφορών. Είναι τεράστια λοιπόν αυτή η συμφωνία με πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα. Δύο θέματα υπάρχουν εδώ. Ένα είναι η πρόσβαση στην αγορά και το άλλο είναι η, ρυθμισμένη συνεργασία. Και τα δύο είναι πολύ σημαντικά γιατί πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε νέες υπηρεσίες στους πολίτες μας, στις επιχειρήσεις μας, να μπορούμε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, να διευκολύνουμε τις μεταφορές και αυτό ε, αποτέλεσε επιτυχία των δύο φάσεων που έχουμε ολοκληρώσει. Πιο σημαντικό όμω από αυτό είναι ότι αυτή η συμφωνία ανοίγει την πόρτα για μια πολύ σημαντική συνεργασία σε τομεί όπου η ΕΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχαν δεσμευτεί να συνεργαστούν στο παρελθόν. Ασφάλεια, α πούμε. Περιβάλλον. Ε, πολιτική ανταγωνισμού. Ε, γνωρίζετε όλοι ότι έχουμε συμμαχίε, διατλαντικέ συμμαχίε ε, αυτό δεν έχει ξανασυμβεί και δεν, έχει, δεν έγινε και ε, έτσι ε, απότομα, ξαφνικά. Έγινε με, με πολύ καλή συνεργασία και των δύο πλευρών. Επίσης, για πρώτη φορά υπάρχουν συγκεκριμένες ε, διατάξεις για κοινωνικά θέματα. Η πρώτη φορά που συμβαίνει σε οποιαδήποτε συμφωνία που αφορά εναερείς μεταφορές. Υπάρχει δέσμευση να εφαρμοστεί η συμφωνία χωρίς να υπονομεύονται τα εργασιακά δικαιώματα. Γι' αυτό την υποστηρίζουν και οι πιλότοι ένθεν και ένθεν του Ατλαντικού. Επίση, πολύ σημαντικέ διατάξει ε, για, το περιβάλλον. Ε, η επίτευξη κοινών προγραμμάτων, ε, έβρεση πρακτικών λύσεων, πιο καθαρέ πτήσει, διαχείριση καλύτερη, δυσυνεργασία στην ΙΚΑΟ. Όλα αυτά είναι πράγματα που δεν έχουν ξαναγίνει σε συμφωνία που αφορά ενέργειε μεταφορέ. Έχουμε επιτύχει σε όλα, όχι. Έχουμε απελευθερώσει πλήρω τις δύο αγορές. Όχι. Γιατί υπάρχουν και όρια στο τι μπορούμε να κάνουμε στον τομέα αυτό. Δεν ήταν δυνατό να απελευθερώσουμε απόλυτα και τον έλεγχο και την ιδιοκτησία και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Η συμφωνία όμως εξακολουθεί να έχει μια διαδικασία που μας βοηθά να πάμε μπροστά. Και οι δύο πλευρές ε, είπαν ότι θα, σταδιακά θα ε, άρουν τα, όλα τα εμπόδια που υπάρχουν και η συμφωνία θα αναθεωρείται ετησίως μέσω της κοινή επιτροπής. Εάν η πρόοδο σε, αυτή την, σε αυτό τομέα είναι πολύ αργή, υπάρχουν μηχανισμοί που μπορούν να ξεκινήσουν να λειτουργούν ε, συμπεριλαμβανομένου και ενό μηχανισμού ε, διαβούλευση σε υψηλό επίπεδο. Αν ε, όμως ε, προχωρήσουμε, αν υπάρξει πρόοδος, τότε θα υπάρξει ενίσχυση ε, και των δικαιωμάτων των επιβατών και θα ανοίξει η, αγορά και σε, η συμφωνία αυτή και σε τρίτε χώρε. Το Ελπίζουμε το Κοινοβούλιο να είναι ικανοποιημένο με αυτά τα θετικά βήματα. Ελπίζουμε να μπορέσετε να δώσετε και εσείς την εγκρίση σας όπως το έκανε και το Συμβούλιο. Γιατί αυτή η συμφωνία προχωρά τη συνεργασία, δίνει άμεσα, άμεσα και, και μελλοντικά ε, δυνατότητες ε, ανάπτυξης και, όπως είπε και ο κύριος Ζασάντα, εξασφαλίζει την, τα ωφέλη της πρώτης φάσης της συμφωνίας. Αν δεν συμφωνήσουμε σε αυτή, την, σε αυτή την δεύτερη φάση, μπορούμε να πάμε στην πρώτη φάση, γιατί υπάρχει και ε, ρήτρα αναστολής. Οπότε δεν χάνουμε τα δικαιώματα που έχουμε επιτύχει στην πρώτη φάση της συμφωνίας. Είναι δυνατόν να κάνουμε κάτι παραπάνω για τον έλεγχο και την ιδιοκτησία. Ίσως να τεθεί ένα τέτοιο ερώτημα. Το, η απάντηση μου είναι ναι. Αλλά εκεί χρειαζόμαστε εσά. Χρειαζόμαστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και χρειάζεται να ε, δημιουργήσουμε ένα διάλογο νομοθετών με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Γι' αυτό η Κομισιόν ε, ε, προτίθεται τον, την άνοιξη του 2011 να κάνει στην Ουάσιγκτον το πρώτο φόρουμ επενδύσεων στις αεροπορικές εταιρείες. Πώς δηλαδή μπορούμε να προσελκύσουμε διεθνή κεφάλαια στον τομέα αυτό. Και θα θέλαμε το Κοινοβούλιο να συμμετάσχει. Γιατί Μόνο μέσω του διαλόγου μεταξύ των νομοθετών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Κογκρέσου να κάνουμε περαιτέρω, να υπάρξει περαιτέρω πρόοδος. Αυτό το θέμα είναι νομοθετικό και για τις δύο πλευρές. Οι διαπραγματευτές ε, έχουν ε, και αυτοί κάποια όρια. Φτάνουν μέχρι το σημείο όταν αρχίζει πλέον να ισχύει η νομοθεσία. Οπότε θα ήθελα να δώσετε και εσείς τη σύμφωνη γνώμη σας, την υποστήριξή σας και νομίζω ότι ε, και τα ενεργά μέλη της Επιτροπής Μεταφορών αλλά και ο Πρόεδρος ε, έχετε πολύ καλές σχέσεις με τους ε, ομολόγους σας στην, στη ΣΥΠΑ και νομίζω ότι είναι ένας τομέας αυτός στον οποίο μπορούμε να συνεργαστούμε. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ κύριε Καγιάκα. Θα πρέπει να φύγω 23 λεπτά για να πάω σε μια συνέντευξη τύπου για τα δικαιώματα των επιβατών Οπότε θα αναλάβει ο Αντιπρόεδρος. Ο κύριος Λάιτφριτ για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κύριε Σιγητά, εξ ονόματος της, ε, του κυρίου Ελ Χαντράουε, σας ευχαριστώ για την εξαιρετική δουλειά που κάνατε. Ο ίδιος βρίσκεται σε μια σημαντική αποστολή στην ε, Πολωνία, οπότε δεν μπορούσε να είναι παρόν, οπότε θα μιλήσω εγώ εξ ονόματός του. Τώρα, Επί αυτή η δεύτερη φάση και η συμφωνία της δεύτερης φάσης είναι ένα βήμα και δεν είναι το τέλος του ταξιδιού. Είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ε, βελτιώνει αρκετά πράγματα, ειδικά για την ε, βιομηχανία την αεροπορική των Ευρωπαϊκών, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αεροπορικής εταιρείας, αλλά σίγουρα δεν είναι το τέλος. Από ό,τι φαίνεται και από τις διαπραγματεύσει δεν, είναι, δεν θεωρούμε ότι είναι πολύ καλό το πώς έχουν τα πράγματα στο θέμα του ανοιχτού ανταγωνισμού ε, μεταξύ, ε, ανάμεσα στον ανοιχτό ανταγωνισμό και την μη ισοσκελισμένη πρόσβαση στην αγορά. Εκεί θεωρούμε ότι η ΕΠΑ έναντι της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πολλά περισσότερα πλεονεκτήματα και οι ευρωπαϊκές ε, αεροπορικέ εταιρείε δεν χάνουν διακριτική μεταχείρισης των Αμερικανικών. Και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Επίση, θεωρούμε ότι η κατάσταση στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε σχέση και με τις ΕΙΠΑ, ειδικά σε ό,τι αφορά τον περιορισμό των, της, ε, της κίνησης, ε, δεν μπορεί να συγκριθεί οι ευρωπαϊκέ μεταφορέ είναι πάρα πολύ πυκνέ, ενώ οι Αμερικανικέ όχι τόσο, οπότε δεν μπορούμε ε, να μιλούμε για τι ίδιε προποθέσει. Και αυτό που αναφέρεται στην ε, έκθεση μέχρι τώρα δεν μπορεί να τύχει της συμφωνή νόμης μας. Θετικό βέβαια είναι ότι υπάρχουν πτυχές κοινωνικές και περιβαλλοντικές. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε ευχαρίστως. Και επίσης η Κοινή Επιτροπή έλαβε ε, υπόψη της και τις πληροφορίες που είχαν δώσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είναι σημαντικό. Για μας, αυτή την, ε, ε, σε αυτή την συμφωνία υπάρχουν θετικά σημεία, βεβαίως δεν έχουμε πετύχει ακόμη τους στόχους που θέλαμε να πετύχουμε. Και στην ομάδα μας, εάν έχουμε συγκεκριμένα δεδομένα και πάει η διαδικασία στην Επιτροπή, θα το συζητήσουμε και θα δούμε αν θα υπερψηφίσουμε ή όχι. Ε, γι' αυτό λέω και πάλι υπάρχουν και θετικά σημεία στην έκθεση, υπάρχουν και αρνητικά. και ακόμη δεν μπορούμε να πούμε ότι φτάσαμε στο τέλος των διπραγματεύσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Καλημέρα σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως ακούσαμε, είμαστε στην δεύτερη φάση αυτού του πρωτοκόλλου που υπεγράφει το Μάρτιο 2010. Και παρά το γεγονός ότι φαίνεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι έχει κάποιες περιορισμένες εξουσίες, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η πραγματική ενημέρωση των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τώρα, πιστεύουμε ότι είναι σημαντική η συμφωνία παρόλα αυτά, δεδομένου ότι η αγορά των αερομεταφορών, των ε, ΙΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το 60% της εναέρειας κυκλοφορίας παγκοσμίω. Άρα είναι υποφελές και για τους δύο. Βεβαίω θα πρέπει να είναι ισοσκελισμένη η συμφωνία αυτή και γι' αυτό θα ήθελα να τονίσω δύο σημεία που κατά την άποψή μου είναι πρωταρχή σημασία και μας απαχωρούν στην ομάδα. Πρώτα απ' όλα, η πρόσβαση θα πρέπει να είναι ισορροπημένη διότι μέχρι σήμερα υπάρχει πραγματική έλλειψη ισορροπίας ε, προς όφελος τον είπα, όσον αφορά τον έλεγχο των αλλοδαπών και την ιδιοκτησία και επίσης θα ήθελα να τονίσω την πρόσβαση αεροπορικών ε, ε, εταιριών που χρηματοδοτούνται. Δεύτερον, το θέμα της βάσης δεδομένων. Πιστεύουμε ότι η βάση δεδομένων θα πρέπει να σέβονται την ιδιωτική ζωή των πολιτών, των ΗΠΑ και της Ευρώπης και πιστεύουμε ότι είναι επίγον να προχωρήσουμε στην θέσπιση κανόνων που θα ισχύουν παγκοσμίω και θα προστατεύουν οπωσδήποτε την ιδιωτική ζωή όλων των πολιτών με εγγύσεις. Τώρα, Τον Ιούνιο του 2010 εγκρίναμε ένα ψήφισμα και πιστεύουμε ότι ο τελικός στόχος αυτών των φωνιών είναι να ανοίξει πλήρως η αγορά χωρίς κανένα περιορισμό. Άρα το τελικό στόχος είναι αυτός. Το γνωρίζουμε. Θα πρέπει να το έχουμε κατά νου και πιστεύω ότι θα πρέπει να ανοίξει και η τρίτη φάση, το συντομότερο δυνατό, για να μπορέσουμε να έχουμε την μεγαλύτερη δυνατή απελευθέρωση, πολύ καλές δυνατότητες εξένες επενδύσεις, βελτίωση των ε, διαφόρων τομέων στους οποίους αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής και να ενισχύσουμε τον συντονισμό ο οποίος όντως ε, προχώρησε τα τελευταία χρόνια αλλά δεν είναι πλήρης. Θα ήθελα λοιπόν να ε, χαιρετήσω την οποιαδήποτε βελτίωση αλλά πιστεύω ότι για να παγιώσουμε αυτή την συμφωνία και τον τελικό μας στόχο να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στα θέματα που μας απασχολούν και τα οποία ανέφερα. Επίσης, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη εκ μέλους της, συναδέλφου Ναταλή Γκρίσμπεργκ, η οποία ε, θα έπρεπε να λάβει το λόγο, αλλά επειδή δεν είναι εδώ, την αντικαθιστώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Μπιλμπάου, κυρία Λιχτινμπέργια. Ευχαριστώ. Πρέπει ειλικρινά να σας πω δεν συμμερίζομαι όλο αυτό το, όλη αυτή την αισιοδοξία για αυτή τη συμφωνία. Ξέρω ότι έχουν εκφράσει και άλλοι τι ανησυχίε τους. Ε, τα πράγματα έχουν ω εξή. Για την πρόσβαση στην αγορά υπάρχουν μόνιμα και ε, μεγάλα προβλήματα για τις ευρωπαϊκές επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή, στη ΣΥΠΑ, που δεν είναι αμοιβαία για μας. Για, δηλαδή, για, για μας υπάρχουν τα προσκόμματα αυτά, για τη ΣΥΠΑ όχι. Δεύτερον, αυτή η κοινή ε, ρύθμιση λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο ώστε οι, οι πάνε πρώτα και μετά εμείς ακολουθούμε από πίσω. Δηλαδή ε, υπάρχει μέχρι στιγμής μεγάλη, ε, μεγάλη διάκριση ίσως να πρέπει να γίνει κάτι από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έναντι των, ε, των ΗΠΑ. Αλλά για την ασφάλεια, για παράδειγμα, από την πλευρά των ΗΠΑ έχουν οριστεί τα πάντα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια για το τι δηλαδή εμείς, ποια είναι τα υπόλοιπα μέτρα πρέπει να πάρουμε για, τον, για την τρομοκρατία, τι θα κάνουμε στο μέλλον. Ε, μάλλον θα πρέπει να στέλνουμε και το βιογραφικό της οικογένειάς μας στο τέλος για να μεταβούμε στη ΣΥΠΑ. Αλλά Υπάρχουν, ε, υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία ακόμα είναι εκρεμή. Για την ασφάλεια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καλούς, καλές ρυθμίσεις, καλές διατάξεις, αλλά δεν έχουμε επηρεάσει τόσο πολύ τα πράγματα τελικά, οπότε εγώ εξακολουθώ να έχω αυτό το πρόβλημα ε, που λέμε συνέχεια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Ε, νομίζω ότι είναι πολύ περιορισμένο ο ρόλος της. Ε, πρέπει πολύ ξεκάθαρα να σας πω ότι ε, υπάρχει τεράστιο περιθώριο για βελτιώσει, γιατί εδώ δεν πρόκειται για ε, μια σχέση ίσου προς ίσον. Μιλούμε για τις παλιές συνήθειες της, του ότι παραβλέπουμε ε, κάποια πράγματα και αυτό πρέπει να σταματήσει. Έχουμε κάποιους θεσμούς κοινού οι οποίοι κάνουν μια πολύ σημαντική δουλειά, συμβάλλουν πολύ σημαντικά, παρόλο που μπορεί καμιά φορά να διαφωνώ με κάποια από αυτά που γίνονται, αλλά πάση περιπτώσει είναι πολύ σημαντική η δουλειά. Αλλά μέχρι στιγμή δεν είδαμε να έχουν αναλάβει κάτι από αυτά που προτείνουμε εμείς οι Αμερικανοί, μόνο το αντίθετο γίνεται. Οπότε δεν υπάρχει ουσιαστική πρόοδος. Αυτό είναι κρίμα. Πολύ κρίμα, γιατί η συνεργασία είναι και σημαντική και σωστή και απαραίτητη. Αλλά για την ε, συνεργασία ε, θα πρέπει αυτό το, αυτούς τους όρους που έχουμε χρησιμοποιήσει θα νομίζω ότι θα πρέπει να τους ε, αφήσουμε. Είναι απλώς έτσι μια θεωρητική αναφορά, δεν είναι καμία δέσμευση αυτή η ρυθμισμένη συνεργασία που λέμε στην έκθεση. Λέμε ναι, αυτά ωραία, με, μεταξύ μας θα το βρούμε, θα συνεργαστούμε για το περιβάλλον, ε, για τα κοινωνικά, αλλά δεν θέτουμε τίποτα για το πώς θα γίνει η μείωση των καυσίμων, ε, για τις νέες μειώσεις επίσης που υπάρχουν ε, τίποτα αυτό δεν έχει προκύψει από την καλή συνεργασία. Εδώ οι ΙΠΑ έχουν, μας έχουν προσπεράσει αρκετά Οπότε νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης για τη σχέση μας με, την, ε, με τη ΣΥΠΑ, πολύ μεγάλο περιθώριο βελτίωσης και νομίζω ότι και η συμφωνία θα πρέπει να ε, ξαναμελετηθεί σε όλες τις, τις λεπτομέρειες γιατί πρέπει να δούμε και τι έχει γίνει από την τελευταία ε, έκθεση και μετά. Εγώ όμως είμαι πάρα πολύ απογοητευμένη πρέπει να σας πω. Αυτή η στρατηγική που ας πούμε ακολουθούμε κι εμείς όταν κάνουν είπα, το πρώτο βήμα, ε, αυτό δεν είναι εκπόνηση πολιτικής, ούτε είμαστε σε μια κατάσταση, σε μια αντιμετώπιση ίσου προς ίσου. Δεν μπορώ λοιπόν εγώ να το δεχτώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γκόρς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι είμαστε σαν να είμαστε σε μια επιτροπή συμφιλίωσης. Μπορεί κανεί να πει ένα ναι ή ένα όχι στο συνολικό πακέτο, να, ζητή να ζυγίσει το ε, βήμα που έχει γίνει προς τα μπρο ή να αμφισβητήσει τα πάντα. Η Κομισιόν είναι αρκετά ε, αισιόδοξη. Δεν θέλω να είμαι ηρωνικός εδώ, αλλά ε, Βλέπω ότι η Κομισιόν δείχνει ότι θέλει να δεσμευτεί, θέλει να προχωρήσει. Βεβαίως, φυσικά δεν έχουμε ε, επιτύχει τους στόχους, ε, προφανώς. Υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες. Ε, στείλαμε μεγάλες αντιπροσωπείες με μεγάλες ε, προσδοκίες και τελικά γυρίσαν πίσω μικρές αντιπροσωπείες με πολύ λίγες προσδοκίες. Δεν θέλω να επαναλάβω τώρα όσα ακούστηκαν, αλλά τα θέματα ανταγωνιστικότητας και περιβάλλοντος είναι σημαντικά, αλλά πρέπει να υπάρξει και μια σύνδεση μεταξύ τους. Δηλαδή αν αύριο ο ανταγωνισμός ε, ε γίνει, ε, προχωρήσει ε, εις βάρος του, των κοινωνικών πτυχών ή του περιβάλλοντος, αυτό δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Και πάλι δεν μπορούμε να τα ακυρώσουμε όλα γιατί μπορεί να ξαναγυρίσουμε στις παλαιές σχέσεις της διμερής των μεμονωμένων χωρών με τη ΣΥΠΑ. Είμαστε σε μια σημαντική χρονική στιγμή και νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ένα βήμα προς τα μπρος. Να συνδέσουμε όμως και το τι γίνεται με την Κομισιόν και το Κοινοβούλιο δεν είμαι εδώ πέρα μόνο για να λέει ένα ναι ή ένα όχι στο τέλος της διαπραγμάτευσης. Ερώτημα λοιπόν δικό μου είναι το η Κομισιόν πώς θα μας εμπλέξει εμάς περισσότερο και πιο ενεργά στην όλη διαδικασία. Εμείς μπορούμε να θέσουμε ερωτήματα. Ε, έχουμε συζητήσει πολλές φορές για τα θέματα αυτά αλλά για τα, στα σημαντικά βήματα φαίνεται ότι το Κοινοβούλιο θα έπρεπε να έχει πολύ πιο ενεργό ρόλο. Αυτό ανεξάρτητα από το μικρό βήμα που θα γίνει προς τα μπρος. Είναι σημαντικό και για εμάς ως Κοινοβούλιο. Είναι σημαντική η συμφωνία αυτή. Να παίξουμε το ρόλο που μας αρμόζει. Να ευχαριστήσω βεβαίως τον εισηγητή και την Κομισιόν και εκ μέρους του ΕΛΚ να πω ότι ε, εμείς θα την υποστηρίξουμε αυτή την ε, πρόταση. Euh, ευχαριστώ. Θα δώσω στον κύριο Καλιέχα και πάλι το λόγο εκ μέρου τη Επιτροπή. Σα ευχαριστώ. Δεν έχω να προσθέσω πολλά πράγματα. Άκουσα αυτή την πολύ ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων ω διαπραγματεύτη, Εγώ εκ μέρου τη Επιτροπής αυτό πέτυχα και σέβομαι τις απόψεις τις οποίες εξέφρασαν οι συναδελφοί σας. Ξέρω ότι ορισμένοι δεν είναι πολύ ικανοποιημένοι και εμείς θα θέλαμε να έχει επιτευχθεί μεγαλύτερη πρόοδος. Πρόκειται για πολύ δύσκολες ε, διαπραγματεύσεις. 7 χρόνια, 9 γύρι, 27 κράτη-μέλη, είπα. Πρέπει να σας πω ότι όλοι όμως ομόφωνα χαιρέτησαν και με θετικό τρόπο και την πρώτη φάση και δεύτερη φάση της συμφωνίας και η αεροπορική βιομηχανία, τα αεροδρόμια, οι ενώσεις πιλότων θεωρούν ότι είναι ένα σημαντικό βήμα προς μελλοντική συνεργασία. Δεν έχουμε φτάσει στο τέλος συνεργασίας. Ανοίγουμε ένα νέο δρόμο για την διατλαντική συνεργασία ένα δρόμο ο οποίος ποτέ δεν είχε μέχρι τώρα ακολουθηθεί στο παρελθόν. οι χώρες δεν θα έχουν με τις ΣΥΠΑ διμερίσια σε θέματα αερομεταφορών. Υπάρχει μία ενιαία συμφωνία η οποία συνάπτεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Υπάρχει μία, ένα θεσμικό όργανο, η Μικτή Επιτροπή, που ενέχεται στις διαπραγματεύσεις, υπάρχουν δυνατότητες συνεργασία σε πολλούς τομείς, ασφαλείας, περιβαλλοντικά, προστασία των καταναλωτών. Έχουμε την δυνατότητα να συζητούμε με τη ΣΥΠΑ νέα μέτρα, ένθεν και ένθεν. Και θα ήθελα να πω στην κυρία Λίχτενμπέργκερ ότι όλα αυτά δεν γίνονται με τρόπο με τον οποίο αυτό θα κάνετε και υπογράψετε και τελείωσε. Και εμεί πολλέ φορέ στάνουμε και του λέμε αυτό πρέπει να γίνει. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στη Μικτή Επιτροπή είναι να βρούμε απόψει ε, στι οποίε θα συμφωνήσουμε και προσπαθούμε να συγκεράσουμε τι απόψει. Ποιο είναι το δικό μας καθήκον, να σεβαστούμε τα προνόμια που έχει ο καθένας και τις προτάσεις του και να βρούμε κοινέ λύσεις αποφεύγοντας αντιφατικές καταστάσεις και δεν θέλουμε να καταστήσουμε ομήρους ούτε τις αεροπορικές εταιρείε ούτε του επιβάτες. Θα προοδεύσουμε διότι έχουμε το πλαίσιο, έχουμε τη Μικτή Επιτροπή και μας διέπουν κοινέ αρχές. Πιστεύω ότι ο τομέας που ανέφερα πολλοί από εσά, δηλαδή η πρόσβαση στις αγορές, όντως είναι ένας τομέας στον οποίο υπάρχουν διαφορετικές θέσεις. Η... Είπα ε, έχουν ανώτατο ποσοστό επειδή 25%, η Ευρώπη 49%. Και είπε ο κύριος ε, πώς μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαδραματίσει ρόλο. Μπορείτε να αλλάξετε την νομοθεσία, μπορείτε να το κάνετε σαν συμφωνήσετε εσείς και το Αμερικανικό Κογκρέσο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί στην επόμενη φάση να δημιουργήσει μία στενή σχέση μεταξύ των δύο νομοθετών. Έτσι μπορείτε κάπως να επηρεάσετε τα πράγματα. Τώρα, για να απαντήσω και στην άλλη ερώτηση του κ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όντως χαιρετίζει σε αυτό το τομέα ένα πιο δυναμικό ενεργό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ελπίζουμε ότι του χρόνου θα μπορέσουμε να οργανώσουμε ένα ε, φόρουμ για θέματα επενδύσεων. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε ειδικού σε θέματα ε, νομοθεσίας και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Ξέρουμε ότι εσείς έχετε μία ε, αποστολή ε, από την οποία θέλετε να αποκομίσετε πολλά. Ε, και εγώ παρόλα αυτά, παρόλα τα προβλήματα σας λέω ότι είμαι αισιόδοξο. πιστεύω ότι υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω πρόβλημα. Ξέρουμε ότι ε, έχουμε, είχαμε ευρωπαϊκές συμμαχίες μέχρι τώρα, τώρα έχουμε συμμαχίες και πέραν του Ατλαντικού, δεδομένου ότι μπορούμε τώρα να συμφωνήσουμε σε θέματα ε, στα οποία οι τρεις ευρωπαϊκές, αν θέλετε, συμμαχίες που έχουμε δημιουργήσει μπορούν να μας ε, φέρουν σε πολύ ισχυρή θέση σε θέματα ε, δικαιωμάτων. Τώρα, μισοάδιο ή μισογεμάτο είναι το ποτήρι. Για ορισμένους δεν είναι αρκετά γεμάτο. Εγώ θα έλεγα ότι αν συνεχίσουμε και προχωρήσει αυτή η συμφωνία, θα μπορέσουμε να ε, συνεχίσουμε να γεμίζουμε περαιτέρω το ποτήρι. Και τελικά φαντάζομαι ότι θα έχουμε την δυνατότητα να έχουμε ε, μία ε, διατλαντική αγορά αρκετά ικανοποιητική. Αλλά εσείς έχετε το τελευταίο λόγο. Και η Κομισιό έχει ολοκληρώσει το έργο της ως ε, θεσμικό όργανο που έκανε την διαπραγμάτευση. Αν δεν σας ικανοποιεί αυτή η συμφωνία, εμεί θα πάμε στη ΣΥΠΑ και θα πούμε, ακούστε, δεν γίνεται αποδεκτή, προχωρήστε λίγο περισσότερο. Πριν να δώσω το λόγο στην εισηγητή. Η κυρία Λίχτενμπέργκερ θέλει να προσθέσει κάτι. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Ένα ερώτημα έχω μόνο. Η ΕΠΑ έχουν λάβει αυτά που θέλανε. Τι κίνητρο έχουν οι ΕΠΑ να πάνε παρακάτω, αφού ό,τι ήθελαν το κέρδισαν. Εμείς θέλουμε τώρα κάτι. Εμείς δώσαμε αυτό που θέλανε οι ΕΠΑ. Οι ΕΠΑ περίπου μας είπανε ναι ίσως μπορεί και εσείς να πάρετε κάτι. Οπότε εμείς σε τι βασίζουμε ακριβώς το ότι η θα προχωρήσει. Αυτό είναι το κίνητρο για το αν είναι το ποτήρι άδειο ή γεμάτο. Εγώ δεν βλέπω ποιο είναι το κίνητρο για τη ΣΥΠΑ να συνεχίσουν να διαπραγματεύονται μαζί μας. Αφού αυτά που θέλανε τα πετύχανε. Ε, αυτό είναι το ουσιώδες για μένα. Εντάξει, μια συμφωνία πάντα είναι μια, ένα βήμα σε μια μακρά διαδικασία. Αλλά σε κάθε βήμα πρέπει να εξασφαλίζουμε ότι και η άλλη πλευρά έχει κάποιο κίνητρο να συνεχίσει να διαπραγματεύεται. Αυτοί έχουν κερδίσει αυτό που θέλανε, το καλάθι τους είναι γεμάτο, εμείς έχουμε έτσι μια, μια σφιχτή χειραψία και μια υπόσχεση. Αν μου πείτε πολύ συγκεκριμένα, εσείς για ποιο λόγο έχετε τόση, είστε τόσο αισιόδοξοι ότι δηλαδή οι ΙΠΑ ακόμη έχουν κίνητρο να συνεχίσουν να διαπραγματεύονται μαζί μας, αλλά συγκεκριμένο απτό κίνητρο, όχι επειδή είμαστε και εμείς καλοί και αυτοί καλοί άνθρωποι, αλλά ε, τότε θα μπορούσα να το σκεφτώ. Αλλά προς το παρόν, έτσι όπως διαβάζω εγώ τη συμφωνία αυτή, η κατάσταση έτσι έχει. Απ' την άλλη μεριά δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνεχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Πήραν αυτό που ήθελαν, τελειώνει εδώ. Μπορείτε να απαντήσετε σε αυτή την ερώτηση. Κάνετε λάθος, κυρία Λίχτεμπεργκεν. Δεν πήρα ότι να είπα. Υπάρχουν ε, πολλά θέματα τα οποία παραμένουν κρεμή και εξαρτώνται από την περαιτέρω πρόεδρο. Δεν ε, μπορούν ε, να ελέγχουν τις ευρωπαϊκές αερογραμμές ούτε να τις αγοράσουν. Δεν έχουν όλα τα δικαιώματα που έχουμε εμεί. Έχουμε αφήσει πράγματα παίξω για να τα διαπραγματευτούμε στο μέλλον. Είναι λαθασμένο να λέγεται πήραν ό,τι ήθελαν και εμείς δεν ε, υλοποίησαμε τους στόχους. Κανένας δεν έχει ε, υλοποιήσει τους τελικούς στόχους διότι δεν έχει πλήρως απελευθερή ώρα. Αλλά για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε πρέπει όπως προβλέπει και η συμφωνία να ε, φτιάξουμε ένα σύστημα. Δεν μπορούν όπως σας είπα να αγοράσουν οι ΙΠΑ. Ε, τις ε, δικές μας ε, αεροπορικές εταιρείες δεν έχει πλήρως απελευθερωθεί η αγορά, δεν έχουν δικαιώματα που έχουμε εμείς. Υπάρχουν δικαιώματα τα οποία θα αποκτήσουν όταν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Μη λέτε λοιπόν, είναι λαθασμένο να λέτε ότι οι μεν τα απέκτησαν όλα και οι άλλοι τα Πρόκειται για μια συνεχή διαδικασία, δεν τελείωσε η διαπραγμάτευση. Κύριε Ζασάντα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την άκρως ενδιαφέρουσα συζήτηση. Το θέμα είναι πολύ επίκαιρο. Το ανέφερα αυτό άλλωστε στην ε, αρχή των συζητήσεων. Δεν ήθελα να δημιουργήσω πρόβλημα όταν έκανα την πρώτη μου παρέμβαση και εξέφρασα κάποιες ανησυχίες. Προφανώς μπορούμε να συζητούμε τα θέματα όπως είναι η μείωση του θορύβου και η ανταλλαγή προσωπικών στοιχείων των επιβατών και το πρόγραμμα Fly America και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι ευρωπαϊκές εταιρείες οι οποίες τώρα δεσμεύονται ως υπεργολάβοι και δεν μπορούν να υπογράφουν οι ίδιες απευθείας ε, συμφωνίες. Πολλά απομένουν να υποθούν για το θέμα και χαίρομαι που υπάρχει προθυμία για συνεργασία. Συνεργασίας μεταξύ των σκιωδών εισηγητών των διαφόρων πολιτικών ομάδων. Και όπως είπα και στην αρχή, η αξία της συμφωνίας είναι η ίδια ύπαρξή της. Αν λέγαμε όχι στη συμφωνία, θα ξεκινούσαμε το μηδέν. Θα πηγαίναμε στην πρώτη μέρα των διαπραγματεύσεων και θα χάναμε πιθανώς πολλά μέχρι τώρα ε, επιτευθέντα αποτελέσματα. Ποια είναι η προσωπική μου άποψη. Πιστεύω ότι αυτό το δεύτερο στάδιο είναι άκρος φιλόδοξο. Πετύχαμε όλους τους στόχους. Όχι θα έλεγα διότι εκκρεμούν πολλά προς επίλυση κατά τον τρίτο γύρο των διαπραγματεύσεων. Και πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει περισσότερο λόγο σχετικά με τα όσα θα γίνουν στον τρίτο γύρο. Οι σημερινές μας λοιπόν ανησυχίες δεν θα μας υποχρεώσουν να καταψηφίσουμε το έγγραφο, διότι επαναλαμβάνω αυτά που προανέφερα. Είναι πολύ σημαντικό το έγγραφο, πραγματικά σημαντικό και θα ήθελα να συστήσω σε όλους να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας στο επεξηγηματικό σημείωμα. Δυστυχώς δεν μπορούμε να υποβάλουμε τροπολογίες, διότι θα έπρεπε κάποια σημεία να τύχουν της προσοχής μας. Τώρα όσον αφορά τις απόψεις που ακούστηκαν, όλες τώρα, κυρίως της κυρίας Μπιλμπάου και της κυρίας Λίχτεμπερ. Και εγώ έχω τις ανησυχίες μου και πολλές ανησυχίες. Θα ήθελα να υπερψηφίσω το έγγραφο παρά τις επιφυλάξεις και ανησυχίες μου. Πιστεύω και θα το ξανασυζητήσουμε αυτό, ότι θα μπορέσουμε να διαλύσουμε τις ανησυχίες που υπάρχουν στον τρίτο γύρο των διαπραγματεύσεων. Αυτά έχω να πω σε αυτή τη φάση. Σας ευχαριστώ όλους για τις απόψεις σας, για τις συστάσεις σας. Θα ήθελα να λάβω υπόψη λοιπόν τα όσα είπατε και τα όσα προτείνατε. Ευχαριστώ κυρία Ζάδα. Καταλάβαμε ότι υπήρχε μια μέρημνα για σημερία και ισορροπία και ελπίζω να υπάρχουν ακόμα πραγματευτικά στοιχεία. Θέλει να, συμμετάσχει, να συμμετάσχει θετικά το Κοινοβούλιο. Θα γίνει ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή προβλέπετε, αλλά ε, έχουμε, μείνει, έχουμε προχωρήσει πιο γρήγορα, δεν ήσασταν αρκετά ομιλητικοί. Περιμένουμε λοιπόν την κυρία Γιούτα Χαουγ που προεδρεύει της Επιτροπής και την κυρία Ποδιέδο που είναι μόνιμη συγκητής για να συζητήσουμε τα στρατηγικά δικηβεύματα όσον αφορά τον προπολογισμό. Στις 10.30 θα το συζητήσουμε το θέμα. Όπως λένε στο στρατό, λοιπόν, μπορείτε να διαλυθείτε για να πάτε για ένα τσιγάρο. Okay, colleagues, um, if I can restart the, the, the meeting. Ας ξεκινήσουμε ξανά τη συνεδρία συνεδρίαση, συνάδελφοι. Έχουμε μέχρι τις 12 ανταλλαγή απόψεων με τους συναδέλφους της ε, Επιτροπής ΣΟΥΡ. Το 13 και το 14 θα το εξετάσουμε μαζί. Ισπανία είναι στο κύκλωμα. Γεια σου Μαδρίτη, εδώ Μαδρίτη. Μαδρίτη ακούτε. Καλώς. Μπορούμε να έχουμε τους, ε, τις ψήφους της ε, Ισπανικής ε, Επιτροπής. Λοιπόν, ε, τα, τα σημεία 13 και 14 μαζί να τα εξετάσουμε. Χαίρομαι όλος ιδιαίτερος που η Γιούτα Χάουγκ είναι εδώ μαζί μας, η πρόεδρος Επιτροπής ΣΟΥΡ. Είμαστε πολύ ευγνώμονες για την παρουσία σας. Και, και που είναι εδώ και ο κύριος Γκαρίγα και διαθέτετε το χρόνο σας να μιλήσετε στην Επιτροπή θα καταλαβαίνετε πόσο σημαντική θεωρούμε την Επιτροπή σας, το ρόλο της και πόσο σημαντική θεωρούμε τη δική μας Επιτροπή. Πάντα θεωρούσαμε ότι η Επιτροπή μας είναι η σημαντικότερη Επιτροπή στον κόσμο. Όχι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόνο, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι χρειάζεται να συνεργαστούμε με άλλες επιτροπές και ιδιαίτερα Γιούτα θέλουμε, επιθυμούμε διακαώς να σε ακούσουμε. Να ακούσουμε εσένα και τους συναδέλφους σου να μας πεις πράγματα για τη δουλειά σου. Θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί σου. Όσο καλύτερα μπορούμε, θέλουμε να δουλέψουμε μαζί σου. Να σου δώσω το λόγο για να ξεκινήσεις. Είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ που και οι δύο διαθέτετε χρόνο να είστε στην Επιτροπή μας. Εγώ ευχαριστώ για την ε, πρόσκληση. Η Επιτροπή Μεταφορών είναι η πιο σημαντική επιτροπή. Χωρίς μεταφορές δεν μπορούμε να πάμε πουθενά μόνο με τα πόδια μας ή με ένα ποδήλατο, αν θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε. Αλλά, ε, και πολύ μακριά δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε με αυτούς τους δύο τρόπους, είναι σίγουρο. Η Επιτροπή μας, να πω κάτι γενικό για την Επιτροπή μας και πώς ακριβώς ε, λειτουργήσαμε, πώς δουλέψαμε και ο κύριος Σαλβαδόρ είναι ο εισηγητής μας ο οποίο μπορεί να μπει σε περισσότερε λεπτομέρειε. Είχαμε την, δημιουργηθήκαμε ως Επιτροπή με την εντολή, από τον, με εντολή από τον Ιούνιο, με, πριν από το καλοκαίρι λοιπόν, πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές ξεκινήσαμε να δουλεύουμε και μετά με, δημιουργήθηκε η Επιτροπή και μετά το καλοκαίρι ξεκινήσαμε να δουλεύουμε. Η πρώτη φάση της δουλειάς μας ε, ολοκληρώνεται σιγά σιγά. Είχαμε κάποιες οριζόντιες πτυχές, ε, ασχοληθήκαμε με οριζόντιες πτυχές της δουλειάς μας. Ε, μιλήσαμε δηλαδή για την ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Ε, συζητήσαμε για την ε, στρατηγική ε, του Ευρώπης 2020. Προσπαθήσαμε να κατανείμουμε λίγο αρμοδιότητες για, τις, ε, για τη δομή των επόμενων δημοσιονομικών προπτικών. Είδαμε τι γίνεται με την εφαρμογή, τι γίνεται με το δημοσιονομικό μας κανονισμό και πώς αυτός έχει αλλάξει. Και χτες και προχτές, Δευτέρα και Τρίτη, κάναμε μία ακρόαση με τέσσερα πάνελ με εμπειρογνώμονες οι οποίοι από απ' έξω μας, μας έδωσαν τη δική τους ε, ε, πτυχή, τη δική τους οπτική γωνία για την στρατηγική για το 2020, για το SMART, που είναι δηλαδή ε, έξυπνη, ε, βιώσιμη και συμπεριληπτική. και ακούσαμε αρκετά προβοκατόρικες σκέψεις, ε, ε, αρκετά πράγματα που είναι λίγο έξω από τη δική μας ε, σκέψη. Ακούσαμε πολιτική συνοχή για τους πιο φτωχούς, γεωργική πολιτική και έρευνα, επενδύσεις στην έρευνα. Και τα υπόλοιπα ας τα αφήσουμε στην άκρη. Εντάξει, αυτό ήταν το πιο επαναστατικό για μένα τουλάχιστον που ακούστηκε. Δεν νομίζω όμως ότι θα εφαρμοστεί κάτι τέτοιο και δεν φαντάζομαι ότι τα κράτη-μέλη θα συμφωνήσουν σε κάτι τέτοιο. Αντί να πιέζουμε έτσι ελαφρώς για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού ε, ε του ευρωπαϊκού πνεύματος ε, να τους αναγκάσουμε είτε μέσω του προπολογισμού είτε μέσω νομοθεσίας να ρυθμίσουν τα, τα του οίκου τους. Κάναμε τη συζήτηση για τον προπολογισμό του 2011 και πώς όλα αυτά ε, συνδέονται, τι γίνεται με τα κρατημέλη, πόσο, πόση πειθό θα χρειαστούμε ακόμη για να τους ε, πείσουμε ότι πρέπει να σκεφτόμαστε όλοι κοινά ευρωπαϊκά. Τώρα, η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει στις 13 Ιανουαρίου. Σας καλώ όλους στην, ε, στις συνεδριάσεις μας. Εκεί θα ασχοληθούμε με τα τομεακά θέματα. Τομεακά σημαίνει θα μιλήσουμε α, ε, για τη γεωργία, για την πολιτική συνοχής, Ε, έρευνα, ανάπτυξη και κάτι που ίσως να ενδιαφέρει τις δικές σας, τη δική σας επιτροπή, τα διευρωπαϊκά δίκτυα, τα TNT. Όταν κλείσουμε αυτή την τομεακή συζήτηση, θα πρέπει να υπάρξει μια έκθεση Ε, εντάξει, το πρέπει, εν πάση περιπτώσει, ακούγεται λίγο υποχρεωτικό, σαν να τον αναγκάζουμε το Σαλβαδόρο να κάνει την έκθεση, αλλά θα πρέπει να προκύψει. Ε, έτσι ώστε το Μάη στην Επιτροπή να μπορέσουμε να ψηφίσουμε την έκθεση και τον Ιούνιο να πάει στην Ολομέλεια και να ζητήσουμε τη στήριξη της Ολομέλειας. Ελπίζουμε να έχουμε τα τρία τέταρτα των ε, ευρωβουλευτών με το, με το μέρος μας ώστε να είναι ισχυρή η θέση του Κοινοβουλίου με τα, με το, στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, να είναι συγκεκριμένη η θέση μας και ελπίζουμε τα τρία τέταρτα των, ευρωπαϊκών, των ευρωβουλευτών να είναι μαζί μας. Αν τα καταφέρουμε τότε θα έχουμε μια σημαντική ισχυρή θέση, θα έχουμε εκπροσώπηση από όλους, βορανό το δύση και ανατολή, θα μπορέσουμε να βουλώσουμε και τα στόματα των ευρωσκεπτικιστών Δεν θέλουμε 90% ή 100% ε, υποστήριξη, αλλά θεωρώ ότι τα 3 τέταρτα των ευρωβουλευτών είναι ένας ε, πολύ ικανοποιητικός αριθμός. Μέθοδος ε, εργασίας. Έχουμε και τις συνεδριάσεις των συντονιστών, αλλά για τη συζήτηση στις ε, συνεδριάσεις της Επιτροπής, ο Σαλβαδόρ ε, προετοιμάζει ένα έγγραφο ε, στοχασμού για, την, για το πώς θα δομήσουμε δηλαδή τις συζητήσεις μας και ο Σαλβαδόρ από τα έγγραφα αυτά θα ε, θα δημιουργήσει και με τη συμβολή των ε, γνώμεων των ε, συναδέλφων τα έγγραφα εργασία. Τα έγγραφα αυτά εργασία δεν είναι επίσημα αποφασισμένα ω κομμάτι τη Επιτροπή, αλλά αυτά τα έγγραφα εργασία θα μπουν στην ιστοσελίδα μα και όποιο ενδιαφέρεται μπορεί να τα μελετήσει. Οπότε αυτή θα είναι έτσι λίγο πολύ μια συμπεφωνημένη εντός της ε, Επιτροπής μας θέση. Είμαστε 50 μέλη στην Επιτροπή μας, 48 ε, αναπληρωτές. Έρχονται πολλοί, ε, πολλά αναπληρωματικά μέλη στις συζητήσεις μας, στις συνεδριάσεις μας. Συζητούμε πολύ, γίνεται ανταλλαγή απόψεων. Επίσης, παράλληλα με τις εργασίες της Κομισιόν, λειτουργούμε κι εμείς, γιατί η Κομισιόν ξέρετε ότι έχει μια task force, μια ομάδα κρούσης, ε, επιτρόπων, η οποία για την Κομισιόν θα προετοιμάσει τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Η Κομισιόν θέλει στο τέλος του Ιουνίου του 2011 αρχέ Ιουλίου να, υποβάλει την πρότασή τη. Αν λοιπόν εμείς θέλουμε να ανταποκριθούμε στις, ε, στις, ε, στη δουλειά μας και να μπορέσουμε να επηρεάσουμε την ε, απόφαση της Κομισιόν με τη δική μα έκθεση, τότε προφανώ θα πρέπει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής που θα ξεκινήσουμε να είμαστε σε επαφή συνέχεια με, το, με την Κομισιόν, να, έχουμε, να κάνουμε κάποιε συζητήσει. Ο επίτροπος που είναι ο σύνδεσμος μεταξύ της Task Force της Κομισιόν και της Επιτροπής SURE είναι ο Γιάννος Λεβαντόφσκι, ο επίτροπος ε, ε, του προπολογισμού. Έλαβε την εντολή από τον ε, από τον παρόσο να είναι ο σύνδεσμός μας και είτε έρχεται αυτό στι συνδετήσεις μας, είτε έρχεται ο Γενικό Διευθυντή τη ε, αντίστοιχης Γενικής Διεύθυνσης που ασχολείται, είτε ο επίφθονο της ε, μονάδας που είναι, που είναι με τον προπολογισμό. Ε, θα βάλω μια τελεία εδώ και ο Σαλβαδόρ ε, θα πάρει το λόγο για να σας πει περισσότερα πράγματα επί της ουσίας. <laughs> Ευχαριστώ πολύ και τους δύο Προέδρους. Ευχαριστώ τους ε, συναδέλφους και την Ντομινίκ που είναι μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμών και είναι ο σύνδεσμος μεταξύ μια τόσο σημαντική επιτροπή που ειδική σε θέματα που αφορούν τις δαπάνες όπως η τρανς και μια τόσο επίσης σημαντική επιτροπή όπως το προπολογισμών. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με δύο σημαντικές, διαφορετικές αλλά λένε μεταξύ τους ε, επιτροπές. Για το θέμα της προετοιμασίας και λειτουργίας της Επιτροπής ΣΟΥΡ δεν έχω να προσθέσω τίποτα περισσότερο. Η Πρόεδρος ήδη εξήγησε τα πάντα, άρα εγώ μπορώ να ασχοληθώ απευθεία με το συγκεκριμένο μας θέμα, που είναι η γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών, του Πρόεδρου Σίμψον συγκεκριμένα. Στην ΣΟΥΡ βρισκόμαστε σε μία προκαταρτική φάση, δηλαδή τα πρώτα έγγραφα ε, τα μελετούμε για να κάνουμε κάποιες κρίσεις, κάποια σχόλια που θα είναι σημαντικές και θα κάνουν τον εισηγητή να αλλάξει άποψη. Αυτό που εμένα με ενδιαφέρει να έχω την μεγαλύτερη δυνατή συνένεση, δεδομένου ότι θα πρέπει να μεταφέρει ένα πολιτικό μήνυμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δηλαδή τα θέματα που αφορούν την προπαρασκευή την επόμενων δημοσιονομικών προοπτικών θα πρέπει να υπάρχει συνένεση και αποδοχή ευρύτερη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όσον αφορά τα θέματα που αφορούν ε, τις μεταφορές. Δεν έχουμε ακόμη ε, μαζί του. Σας ευχαριστώ διότι μας επιτρέπετε με αυτή τη συνάντηση να δούμε ποια είναι τα προβλήματα που σας απασχολούν βάσει της εμπειρίας την οποία έχετε εσείς κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου προγραμματισμού και ποια είναι τα θέματα που πιστεύετε ότι θα είναι σημαντικά στο μέλλον. Ακόμη δεν ξέρουμε στην ΣΟΥΡ και ποια θα είναι η μελλοντική δομή των ε, δημοσιονομικών, ε, δημοσιονομικών προοπτικών και πού θα πρέπει να μπει το κομμάτι το οποίο αφορά ε, Δεν ξέρουμε δηλαδή πώς θα δομηθεί. Θα πρέπει να έχουμε πολύ μία δομή ε, στην οποία θα έχουμε πολύ λίγες ε, ε, κεντρικές γραμμές πλεύσεως ή θα πρέπει να κάνουμε κάτι το διαφορετικό από τα πλαίσια της στρατηγικής 2020. Πρέπει να σας πω ότι και εμείς και η πρόεδρος, πρόεδρος θέλουμε να μιλήσουμε με και δεν ξέρουμε ακόμη ποια θα είναι η σχέση μεταξύ της στρατηγικής 2020 και των μελλοντικών δημοσιονομικών προοπτικών. Όπως πάντα, οι ιδέες και τα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ασαφείς και δεν μπορούμε εμείς στην πράξη να τα μεταφράσουμε για να δούμε τι σημαίνει αυτό για τον προϋπολογισμό τα επόμενα 5, 6, 7, 10 χρόνια. Ίσως θα έχουμε λοιπόν μία δομή πιο περιορισμένη, αλλά αυτό το οποίο θα πρέπει να δούμε είναι να δούμε πώς δομείται πάνω εδώ η πολιτική των μεταφορών. Διότι όπως λέτε και εσείς στην εκθεσή σας, πρόκειται για μία από αυτές τις ε, ε, επιτροπές που προσδίδει μεγάλη προστιθέμενη αξία στον προϋπολογισμό. Σε αυτές λοιπόν τις υποδείξεις που μας κάνετε, Μπορώ να πω ότι συμφωνούμε με πολλές. Όπως ξέρετε, ένα από τα πρώτα πράγματα τα οποία μπορέσαμε να ανοιχνεύσουμε στις παρούσες δημοσιονομικές προοπτικές είναι ότι υπήρχαν ελάχιστα κονδύλια για τα διευρωπαϊκά δίκτυα των μεταφορών. Αυτό νομίζω ότι είναι λανθασμένο, γι' αυτό δημιούργησε και διάφορα οικονομικούς στραγγαλισμούς και προβλήματα και δυσχεραίνει την ανάπτυξη των ε, μεγάλων δικτύων τα οποία και στο παρελθόν αλλά και τώρα είναι πρωταρχική σημασία για την εξέλιξη της Ευρώπης. Ούτως ή άλλως, στα έγγραφα τα οποία εκπονούμε στην Επιτροπή μας, το πιο σαφές παράδειγμα προστέμενης αξίας. Έχουμε δύο συγκεκριμένα που μας αποδεικνύουν ότι μια κοινοτική πολιτική μπορεί να έχει προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκή κλίμακα, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την χορήγηση των πόρων. Πρώτα απ' όλα, πρόκειται για τις δαπάνες που προβλέπονται για την έρευνα και την ανάπτυξη και δεύτερον αυτά κονδύλια τα οποία θα δοθούν για την ανάπτυξη των έργων υποδομής στον τομέα των μεταφορών. Είναι λοιπόν ε, σαφές ότι η μεταφορά ε, ότι αν, δεν υπάρχ, ότι αν υπάρχουν αρκετά κονδύλια και στους κρατικούς προϋπολογισμούς και στον κοινοτικό για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν έργα υποδομής στον τομέα των μεταφορών είναι κάτι το οποίο είναι γενικότερα πολύ επωφελές. Συμφωνούμε λοιπόν με το σημείο 6 και με το σημείο 7 που είναι ένα από τα βασικά θέματα για τις μελλοντικές δημοσιονομικές προοπτικές. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατή χρηματοδότηση των διευρωπαϊκών δικτύων στον τομέα των μεταφορών. Στο σημείο 8 επίσης αναφέρεται τη στρατηγική 2020 Αναφέρεται λοιπόν με σαφήνεια ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει ε, ικανοποιητική χρηματοδότηση αυτών των δικτύων. Βεβαίως θα συζητήσουμε το όλο θέμα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που μεταξύ άλλων είναι από τους μεγάλους φορείς χρηματοδότησης. Στο σημείο 9 έχουμε ένα σημείο που είναι σύνηθες μεταξύ όλων των επιτροπών, δηλαδή ζητούμε αύξηση της χρηματοδότησης για τα δέθων μεταφορών. Αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο θα το ζητήσουν και άλλες επιτροπές. Αναφέρεστε επίσης στην ε, δυνατότητα ενδεχομένως κάποιοι πόροι για τη συνοχή να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν και έργα μεταφορών. και βεβαίως αναφέρεστε στην ε, κοινοτική χρηματοδότηση για τα ΔΕΔ, ενώ από τους κρατικούς προπολογισμούς θα πρέπει να δίδονται πόροι για τα κεντρικά δίκτυα των ΔΕΔ. Πρέπει να σας πω ότι για το 2007-2008, ήδη έχουν δεσμευθεί όλα τα ποσά που αφορούν τα δέδια της μεταφορές. Βεβαίως γνωρίζουμε ότι ήταν απαραίτητο να γίνουν τέτοιο, αλλά ξέρουμε ότι είναι ανεπαρκή τα κονδύλια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το πούμε στις παρατηρήσεις μας. Το Γαλιλαίο και το Μάρκο Πόλο είναι προγράμματα μίζωνος στρατηγικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι σημαντικό διότι ζητείται και αύξηση των πόρων για τον Γαλλία. Δυστυχώς, δεδομένου ότι η χρηματοδότηση του προκοινωτικού προπολογισμού δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε, χρειάστηκε να μεταφέρουμε κονδύλια από τη Γεωργία για να χρηματοδοτήσουμε τον Γαλιλαίο. Αυτή η πρακτική δεν μας αρέσει καθόλου, διότι ε, αυτό το οποίο κάνει είναι να παρουσιάσει μία λανθασμένη εικόνα των πραγμάτων, αλλά ξέρουμε ότι εδώ έχουμε συγκεκριμένη περίπτωση να κάνουμε με σχέδια, με προγράμματα τα οποία πραγματικά προσφέρουν προστιθέμενη αξία στον κοινοτικό προπολογισμό. Τα θεωρούμε λοιπόν πολύ σημαντικά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για τις προτάσεις σας θα τις χρησιμοποιήσουμε όταν θα μελετήσουμε την μελλοντική δομή των ε, ε, δημοσιονομικών ε, πρόπτικων και όταν θα κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις, αλλά πρέπει να σας πω ότι τα δέδη των μεταφορών θα πρέπει να εξετάζονται από την πρίσμα της ειδική προστιθέμενης αξίας για όλη την Ευρώπη. Και αυτό να ληφθεί υπόψη όταν θα γίνει ο υπολογισμός των κονδυλίων που θα δοθούν σε εσά. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, Σαλβαδόρ. Να κάνω εισαγωγή στην έκθεσή μου της. Διότι εξετάσουμε και τις δύο μαζί και θα μιλήσουμε μετά τα μέλη τα μέλη αυτής της Επιτροπής είναι οι δικοί τους τομείς τους. Ενθαρρύνθηκα από αυτά που άκουσα να λες όσον αφορά την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Αυτή θα είναι μια από τις προτεραιότητες που θα θέσουμε όσον αφορά το TEN-T. Θα είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σου. Βαρέθηκα αυτό το δίκτυο TEN-T που είναι με προγράμματα 27 κρατών μελών τα οποία δεν συνδέονται μεταξύ τους. Αυτό που θα κάνουμε είναι η διασυνοριακή πτυχή να αποκτήσει προτεραιότητα, να διασυνδέσουμε αυτά που ήδη έχουμε. Η κυρία Γιάλα Σέντερ θα μιλάει επί ώρες για το Περπινιό Βαρκελόνη και εγώ. Αυτό είναι απλώς ένα παράδειγμα Ξέρουμε ότι σημειώνουμε πρόοδο όταν, θα σημειώσαμε πρόοδο όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση. Ξέρουμε ότι θα φτάσουμε στον δρόμο για τη Δαμασκό, όπως λένε. Χαίρομαι με αυτά που άκουσα λοιπόν, είναι ενδιαφέρον, ε, διότι οι μεταφορές για την οικονομία της Ευρώπης είναι πάνω από 4,5%, 4,6% του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι οι μεταφορές. Και πιστεύουμε, και το λέγαμε αυτό, ότι ένα σύστημα βιώσιμο των μεταφορών ζωτική σημασία για το μέλλον τη Ευρώπη και για το οικονομικό μέλλον της Ευρώπης και για το κοινωνικό και για τη βιωσιμότητα. What you said this morning is... Αυτά που λέγατε το πρωί είναι άκρο ενθαρρυντικά. Δηλαδή κινούμαστε προς την ίδια κατεύθυνση. Πιστεύουμε ότι χρειάζεται καλύτερο συντονισμό των TNT και του Ταμείου Συνοχής. Όταν λέω τέτοια πράγματα, η Επιτροπή Περιφερειακών Υποθέσεων αρχίζει και ανησυχεί. Γιατί θεωρεί ότι ξεκινώ μία επιδρομή κατά των πόρων τους. Δεν πρόκειται περί αυτού. Προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τα, το Ταμείο Συνοχής και τα άλλα θετικά ταμεία στα ευρωπαϊκά πλαίσια και εμείς σαν Επιτροπή Μεταφορών κοιτάμε τι μπορούμε να κάνουμε για να συμβάλλουμε. Αρχίζουμε να συναντόμαστε και με τα μέλη της Επιτροπής Περιφερειακών Υποθέσεων στην ομάδα μας για να τους καθησυχάσουμε. Ότι δεν είμαστε ο Cassidy και ο Sundance Kid, δεν είμαστε ληστές, προσπαθούμε να τους κλέψουμε. Καμιά φορά έτσι μας βλέπουν. Αλλά υπάρχει περιθώριο να αυξηθούν οι πόροι του Ταμείου Συνοχής που διατίθεται για τις μεταφορές. Και πρέπει να είμαστε ευφυείς και στους άλλους τομείς. Έχουμε το πρόβλημα της αστικής συμφόρησης. Η αστική συμφόρηση δεν περιορίζεται μόνο στην Ανατολική Ευρώπη, στα νέα κράτη-μέλη. Δεν ξέρω πότε θα σταματήσουμε τα λέμε νέα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να είναι 50 χρόνια μέλη για να μην λέμε νέα κράτη-μέλη. Το νέα Ξέρετε όμως θέλω να πω ότι η συμφόρηση η αστική είναι ένα πρόβλημα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρέπει να δούμε πώς μπορούμε αυτό να το λύσουμε μέσω άλλων διαθωτικών ε, πόρων, όχι μόνο από το Ταμείο Συνοχής. Ανέφερε τον Γαλιλαίο. Ο Γαλιλαίος γεννήθηκε κατά κάποιο τρόπο σε αυτήν την Επιτροπή, αλλά έφυγε από το σπίτι και πήγε στην Επιτροπή βιομηχανία. Δεν χαρήκαμε, αλλά αυτή είναι η απόφαση τη. Ε, Επιτροπής της Ευρωπαϊκής μας το επέβαλε. ο ουρανούς, Σίζαρ, όλα αυτά προσπαθούν να δώσουν ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Σωστά την ανέφερες. Κοστίζει, κοστίζει. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα. Πρέπει να δούμε να συνεργαστούμε με τον ιδιωτικό τομέα, τι κυβερνήσει κλπ. για τη χρηματοδότηση όλων αυτών που θέλουμε να κάνουμε. Μάρκο Πόλο, το ανέφερε και αυτό. Τουρισμό τώρα. Είναι η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού εδώ. Μέσω συνθήκης τη Αβώνας που δίνει εξουσία στο κοινοβούλιο, στον τομέα του τουρισμού, έχει αυξηθεί η σημασία μα λόγω του τουρισμού, αλλά δεν υπάρχει κονδύλι. Μηδέν. Μηδέν. Τίποτα. Νάδα για τον τουρισμό. Τι προσπαθούμε να κάνουμε. Έχουμε την παράγραφο 16 του σχεδίου εκθεσής μου. Εκεί αντικατοπτρίζεται το τι μπορεί να κάνει ο τουρισμός. Είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ο τουρισμός και η δυνατότητα οικονομικής ανάπτυξης μέσω τουρισμού ε, είναι τεράστιο. Δεν αφορά χώρες όπως είναι η δική σας και τη Μεσόγειο. Είναι πώς να αναπτύξουμε άλλες περιοχές. Κάποιος μπορεί να αναφερθεί ε, στην πόλη του διότι είναι η πηγή της βιομηχανικής ε, επανάστασης. Ε, και πώς μπορούμε να αναπτύξουμε το βιομηχανικό του ΣΥΠΗΝ ε, τουρισμό, πώς ε, το βιώσιμο τουρισμό, να εκμεταλλευτούμε την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης. Προσπαθήσαμε φέτος να κάνουμε κάτι με τα κονδύλια, δεν ήταν καλύτερη χρονιά, ο Ντομινίκαν έκανε ό,τι μπορούσε. Αλλά όπως είπε και ο Άρνολτ Βαντζενέγκερ, θα ξαναγυρίσω, θα ξαναγυρίσουμε. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε κάποια χρήματα λοιπόν στον τουρισμό, στο εγγύς μέλλον. ενθαρρύνθηκα, αναθάρισα από αυτά που άκουσα. Γιατί είναι καλός ιονός. Δείχνει ότι μπορούμε να συνεργαστούμε. Δεν είναι ότι εμείς θέλουμε να μας δώσετε τα πάντα. Και να δούμε τι μπορούμε να προσφέρουμε και εμείς εσάς. Και εσείς πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε για να περάσουμε αυτή την εικόνα στην Ευρώπη και να ακουστεί η φωνή των μεταφορών. Όπως κάθε άλλη επιτροπή μας αρέσει να μας αγαπούν. Θέλουμε να μας αγαπούν τα μέλη τη Επιτροπή ΣΟΥΡ. Μάθιος για το ΕΛΚΟ, ο κ. Γκόσου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ τους δύο συναδέλφους για την εισαγωγή. Είναι πολύ ενθαρρυντικά αυτά που ακούσαμε, ειδικά κοιτώντα και το τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν πραγματικά πολύ, με, πολύ σημαντική η πρωτοβουλία αυτή να γνωρίσουμε αυτή την Επιτροπή και να οικειοποιηθούμε με, τα, με το αντικείμενό της. Αν μπορέσουμε να υπολογίσουμε και τα δύο από κοινού, 20% του ΑΕΠ της Ευρώπης και περίπου 18, μιλάμε για 20% του ΑΕΠ και 18 εκατομμύρια ε, ε, ε, εργαζομένων στον τουρισμό. Ε, δεν υπάρχει άλλος τομέας που να δείχνει με αποδείξεις ότι όντως έχει μεγάλο δυναμικό όπως αυτός. Βεβαίω έχει και τι αρνητικέ του επιπτώσει, ε, όπω το λέει και ο συνάδελφο Μίχαελ, όχι μόνο στο περιβάλλον. Φυσικά, όταν κάποιο είναι ενεργό, καταναλώνει κιόλα. Προφανώ. Ε, γι' αυτό εδώ για κάποια χρόνια εμεί είμαστε πολύ ενεργοί ώστε να μπορέσουμε να ε, απαλείψουμε αυτέ τι αρνητικέ συνέπειε. Ο τομέα αυτό είναι ένα ε, σημαντικό τομέα που είναι και για την, για την καρδιά τη Ευρώπη. Χωρί ε, μεταφορές, χωρίς τουρισμό, αλλά κυρίως χωρίς, μετα... χωρίς μεταφορές δεν θα είχε ανοίξει η αγορά, δεν θα είχε αυξηθεί η κινητικότητα των πολιτών. Αυτό σημαίνει ότι προφανώς έχουμε στα χέρια μας εδώ με τα TNT ένα πολύ σημαντικό φάκελο. Την τελευταία περίοδο από τις ε, εκλογέ έχουμε ε, δραστηριοποιηθεί πάρα πολύ με, τις, ε, με το περιβάλλον. Όχι μόνο ε, για προγράμματα σε διάφορες χώρες, αλλά και για την ασφάλεια, για τη ρύθμιση των αγορών, για το άνοιγμα των αγορών. Έχουμε θέσει πρότυπα και κοινωνικά. Η πρόσβαση στην αγορά εργασία είναι ρυθμίζεται τόσο πολύ, σε κανέναν άλλο τομέα δεν ρυθμίζεται τόσο πολύ όσο στι μεταφορέ. Έχουμε θέσει λοιπόν κάποιου συγκεκριμένου στόχου. Οπότε νομίζω ότι είμαστε σε έναν, βρισκόμαστε σε έναν τομέα ο οποίο κατά την άποψή μα ε, ξαφνικά έχει ανακαλυφθεί από άλλε επιτροπέ και γι' αυτό δραστηριοποιούνται. Ε, γι' αυτό η στρατηγική 2020 είναι πολύ σημαντική. Η κοινοτομία για μα είναι ένα όρο πολύ σημαντικό, ένα όρο κλειδί για το μέλλον. Η βιωσιμότητα επίση οι κοινωνικές πτυχές. Επίσης, είναι οι τρεις βασικές πτυχές ε, που βρίσκονται εδώ, οπότε δεν χρειάζεται να ψάχνουμε τίποτα άλλο για να κάνουμε τη δουλειά μας και ελπίζω ότι μέσω της δικής σας εργασίας αυτά τα βασικά θέματα που διαπραγματευόμαστε εδώ στην Επιτροπή θα μπορέσουν να δημοσιευθούν ακόμη περισσότερο προς τα έξω, ακόμη καλύτερα. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, αν θέλουμε να ορίσουμε το μέλλον, πρέπει να θέσουμε προτεραιότητες, πρέπει να καθορίσουμε προϋποθέσεις, πρέπει να βελτιώσουμε το συντονισμό. Δεν έχω την ψευδέστηση ότι θα έχουμε περισσότερα χρήματα στο μέλλον. Είμαι μάλιστα πεπισμένος ότι θα πρέπει να, να, να δουλέψουμε καλύτερα με λιγότερα χρήματα. Για να πετύχουμε τους στόχους μας, λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να έχουμε ενισχυμένο συντονισμό σε όλους τους τομείς είτε επιλέξουμε την πρώτη επιλογή είτε τη δεύτερη, ε, δεν είναι το σημαντικό αυτό. Καλό θα ήταν να μην παραμείνουμε στα παλιά, να έχουμε μια νέα προσέγγιση, να μπορέσουμε να προτείνουμε κάτι καινούργιο. Και ακριβώς αυτή η συζήτηση για τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαμε να τη συνδέσουμε με, την, ε, με τα δημοσιονομικά. Οι μεταφορές επίσης θα μπορούσαν να πέσουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Γιατί για μας η συνεργασία με την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι πολύ σημαντική όχι όπως παλιά, αλλά αν διαπιστώνουμε ότι το Ταμείο Συνοχής είναι ένα τέταρτο, δίνει ένα τέταρτο των, ε, των κορδιλίων στην, ε, στις μεταφορές, τότε θα μπορέσουμε αυτό να το χρησιμοποιήσουμε, να το, ε, να το καλλιεργήσουμε, ώστε και ε, ότι, ε, ώστε αυτά τα κονδύλια να πάνε ε, σε επενδύσει, να πάνε σε διευρωπαϊκά δίκτυα, σε διαλειτουργικότητα αυτών. Οπότε πρέπει να συνδέσουμε τον ε, συντονισμό το δικό μα και με άλλε επιτροπέ. Και αυτό ισχύει και για το περιβάλλον. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να, να συζητήσουμε παράλληλα και να δαπανούμε τις δυνάμει μα και, στις, και, στις, και στην έρευνα και, στην, και στις υπόλοιπες συζητήσεις. Νομίζω ότι πρέπει να τα συγκεράσουμε όλα αυτά, να συνδυάσουμε τις προσπάθειές Και βεβαίως πρέπει να συνδέσουμε τις προσπάθειές μας και με άλλες επίρους. Πρέπει να μιλήσουμε με μία φωνή, ειδικά για τον τομέα του περιβάλλοντος, ε, όχι με 27 ξεχωριστέ φωνές. Ένα τελευταίο, Θα έχουμε νέα έσοδα. Θα έχουμε νέους πόρους. Οι ε, μεταφορές ε, θα είναι σαν να τις, ε, να τις συζητούμε για πρώτη φορά πάλι σε λίγο καιρό. Γιατί τα κράτη-μέλη θα διαπιστώσουν ότι ε, δεν θα υπάρξουν νέες, νέες πηγές χρηματοδότησης. Αλλά τουλάχιστον εφόσον υπάρχουν κονδύλια για το τομέα των μεταφορών, ας ενισχυθούν οι, οι, ας τομείς που άπτονται των μεταφορών. Υπάρχουν δύο συνέπειες εδώ. Στα πλαίσια της συζήτησης και των ε, δημοσιονομικών πτυχών, θα πρέπει να δούμε το θέμα του earmarking, της κατανομής των κονδυλίων. Και δεύτερον, αν αύριο μιλήσουμε για προγράμματα PPP, θα πρέπει να προχωρήσουμε ρεαλιστικά με τους ε, ιδιώτες να τους, δω, να τους δίνουμε την ε, δυνατότητα, να, την ε, ευκαιρία να επενδύουν, να τους πούμε ότι εδώ αξίζει τον κόπο να επενδύσετε, γιατί είναι ένας τομέας που θα συνεχίσουμε να το χρησιμοποιούμε. Αυτά τα προγράμματα λοιπόν, τα ΣΔΙΤ ουσιαστικά, είναι ε, ουσιώδους σημασίας. Θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν και, αυτά, και κυρίως στον τομέα των μεταφορών. Είναι πολύ, μπορούμε να βρούμε πολύ ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις για να ενισχύσουμε τα ΣΔΙΤ. Καλύτερες, ε, καλύτερη θέση λοιπόν προτεραιοτήτων, συντονισμός με, άλλες, με άλλους τομείς και αιρεσιμότητα. Να έχουμε δηλαδή κάποια κονδύλια τα οποία να δίδονται στοχευμένα, όχι για την οποιαδήποτε δραστηριότητα. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ κυρία Γιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω πάρα πολύ και την κυρία Χάου και τον κύριο Γκαρίδε Πολιέδα για την ε, παρουσία τους και διότι μας εξήγησαν αυτά τα θέματα. Ξέρουν πόσο σημαντικό είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι δημοσιονομικές προοπτικές και σίγουρα διότι προετοιμάζουν πάρα πολύ καλά αυτή τον αγώνα που πρέπει να κάνουμε κάθε 7 χρόνια. Και βεβαίω αυτό που θέλουμε όλοι βεβαίω είναι για όλου του πολίτε να υπάρχει αυτό που κάνουμε πάρα πολύ μεγάλη προσθέμενη για του πολίτε. Φέτο, πραγματικά πρέπει να πω ότι είμαι πολύ απογοητευμένη. Βλέπω τον συνάδελφο Κρός, ακούω την Κομισιό ε, τι έχει να πει για να μπορέσει να υπάρξει Προπολογισμό. Το πολεμήσαμε, αλλά δεν κατορθώσαμε τίποτε, διότι νομίζω ότι το θέμα τη καινοτομία είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για τι προοπτικέ. ε, λοιπόν, τις επόμενες θα κάνουμε. Οι παρουσες προπτικές... προοπτικές 7-13 ήταν αυτό του ποιοτικού έλματος. αλλά νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε έκκληση στην ε, καλή θέληση όλων και να ακούσουμε αυτά το οποίο είπαν οι συνάδελφοι. Πιστεύω ότι το νέο στάδιο μετά το 2013 θα πρέπει να είναι η στιγμή της ευρωπαϊκής κινητικότητας. Ξέρουμε ότι πολλοί άλλοι πρωταγωνιστές σημαντικοί στον ε, κόσμο, οι τι κάνουνε σε αυτό το τομέα. Και Ξέρουμε πόσο τα έργα υποδομών είναι σημαντικά. Τι κάνουν και η Αφρική και η Λατινική Αμερική. Αν λοιπόν πραγματικά αυτή τη στιγμή και άλλες, άλλοι μεγάλοι ε, ανά τον κόσμο Αυτού τους τομεί θέλουν να ενισχύσουν τη στιγμή που δερχόμαστε μια μεγάλη οικονομική κρίση. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να καθυστερήσει η Ευρώπη και κυρίως να δώσει το μεγάλο πολιτικό μήνυμα ότι για να υπάρχει καλύτερη δυνατότητα κίνηση στην Ευρώπη, καλύτερη κινητό, θα πρέπει να, οθείς, να, να προωθήσουμε τι πολιτικέ που θα δώσουν μεγάλη όθηση στι υποδομέ. Και είναι οι υποδομέ των μεταφορών πολύ σημαντικοί. Βλέπουμε τι συμβαίνει όταν ε, δημιουργείται πρόβλημα. Τι συνέβη από μερικού μήνε το θυμάστε με τι ενέργειε μεταφορέ. Δεν μπορούν ε, οι επίγειες μεταφορέ ε, να αντικαταστήσουν τι ενέργειε μεταφορέ. Γι' αυτό θα πρέπει εμεί να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τι ενισχύσουμε και κυρίω τι επίγειε, τα δικά μα δίκτυα και τι σειροδρομικές. Όπω είπαν πολύ σωστά λοιπόν οι συνάδελφοι, το στίχημα για τους σειροδρόμους δεν σημαίνει μόνο έργα υποδομής, δηλαδή ε, ανοξίδωτο ατσάλι και τσιμέντο, φίρδιν μίγδιν, ασφάλεια για τους πολίτες κυρίως. Πρέπει λοιπόν να μπορούμε να έχουμε τεχνολογία εχμής σε όλη την Ευρώπη. Και όπως ελέγχθη, η προώθηση όλων των ε, ε, ειδών ε, πηγείων μεταφορών, οδικών και σιδηροδρομικών μεταξύ άλλων, είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα βοηθήσει την Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν να δώσει αυτό το πολιτικό μήνυμα, επαναλαμβάνω, η Ευρώπη. Περισσότερες επενδύσει, περισσότερες θέσει απασχόληση, ανταγωνιστικότητα ε, και βεβαίως πρέπει να πω ότι και η ασφάλεια των μεταφορών αυτών, κυρίως των σιδηροδρομικών, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν και άλλα προγράμματα τα οποία είναι και σχέδια πολύ σημαντικά. Ε, το θέμα των ε, εισιτηρίων και πώς εκδίδονται. Ο κατακαιρματισμός των συστημάτων είναι μια μεγάλη αδυναμία. Εν πάση περιπτώσει, κάτι πρέπει να κάνουμε. Αλλά επαναλαμβάνω, το πιο σημαντικό θέμα είναι να δοθεί το πολιτικό μήνυμα για επενδύσεις στην Ευρώπη. Διαφορετικά θα καθυστερήσουμε, θα είμαστε οι τελευταίοι σε αυτό τον αγώνα και θα μας προσπεράσουν οι Άπωνες, οι Κινέζοι, οι Αμερικάνοι και όλοι οι άλλοι. Ο κύριος Γκρίμπα Πολιέδο μίλησε πολύ σωστά για την δυνατότητα που υπάρχει για να μας ε, βοηθήσει και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Όταν μιλούμε για τέτοια θέματα, μιλούμε για ποιος μπορεί να μας βοηθήσει, βγάζοντας εμείς τον εαυτό μας από την ουρά μας από τη μέση. Εγώ πιστεύω ότι εάν αυτή η προσπάθεια σημαίνει ε, προστιθέμενη αξία για την Ευρώπη, ο κοινοτικός προϋπολογισμός θα πρέπει επίσης να βάλει το χέρι στην τσέπη. Γιατί αυτό είναι σημαντικό για τους πολίτες. Επίσης, ε, τα κομβικά ε, σημεία μεταξύ των διαφόρων δεύτερες μεταφορές είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει ασφάλεια και σαφή μηνύματα σας Επίσης, τώρα, το να δώσουν ε, για τις ε, μεταφορές από τα ταμεία συνοχής και από τα διαδικά κάποιους πόρους, νομίζω ότι είναι κάποιο προβληματικό. Καταρχάς, κάναμε κάτι για να μπορέσουμε ε, στις πρώτες φάσεις να καθορίσουμε τις προτεραιότητες για να χορηγήσουμε κονδύλια. Αλλά εγώ πιστεύω ότι η Επιτροπή η δική μας με την συνδρομή των μελών της Επιτροπής ΣΟΥΡΕ θα πρέπει να κάνουμε κάτι ώστε να μπορέσει ο προπολογισμό στα πλαίσια των δημοσιονομικών προοπτικών από το 2014 και μετά να δώσει αυτό το περίφημο πολιτικό μήνυμα σινιάλο προ όλου. Που θα είναι αποφελέ για όλου του Ευρώπη. Και οι υπόλοιποι θα ακολουθήσουν. Δεν μπορεί κανεί να πει ε, όχι σε κοινοτικέ επενδύσει και να περιμένει να έρθουν οι άλλοι να βοηθήσουν. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ. Χαίρομαι που είναι εδώ τα μέλη της ε, Επιτροπής ΣΟΡ. Φυσικά είναι σημαντικές μεταφορές, αλλιώς δεν θα ήμασταν εδώ. Θέλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πέρα από όλα τα υπόλοιπα που είναι σωστά, να αντιμετωπίσουμε και την κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή δεν θα αντιμετωπιστεί αν δεν αλλάξουμε την κινητικότητα. Οι μεταφορές είναι υπεύθυνε για το 30% των εκπομπών αερίων και έχει αυξηθεί από το 90% κατά 35% ε, λόγω της ε, υπερθέρμανσης των κτηρίων, των συστημάτων. Μέχρι στιγμής έχουμε επιτύχει μία, μία μείωση του 10%. Πρέπει λοιπόν να, να συνεχίσουμε να προχωρούμε. Και πρέπει το ερώτημα που, που θα θέσουμε να είναι μετά από 20 χρόνια ε, διευρωπαϊκών δικτύων μπορούμε να προχωρήσουμε, να συνεχίσουμε έτσι. Και αν δεν καταλήξουμε πουθενά, τι θα γίνει. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε θέσει λάθο προτεραιότητε ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χθε είπαμε ότι, στην, ε, ότι το, το Βερολίνο, το Παρίσι-Βερολίνο, Πρατισλάβα δεν είναι ευρωπαϊκό δίκτυο. Είναι ε, εθνικό ουσιαστικά πρόγραμμα που συνδέει του σιδηροδρόμου των χωρών αυτών. Ναι, αλλά εμεί το κέντρο βάρου που θα το θέσουμε. Το κέντρο βάρου τα τελευταία χρόνια θα μπορούσε να πει κανεί είναι μια συλλογή των εθνικών εγωισμών. Κάθε χώρα ήθελε να μπει και να, να συμβάλλει, αλλά όταν μιλούσαμε για τη χρηματοδότηση, κάναν όλοι πίσω. Ιταλία σε τρία μεγάλα, τέσσερα μεγάλα προγράμματα από τα 30. Σε, τέσσερα, σε τρία προγράμματα έχει συμβάλει η Ιταλία, χωρίς όμως να έχει κάνει οποιαδήποτε συμφωνία α, οικονομική. Γι' αυτό όταν ε, οργανώνουμε τέτοια προγράμματα πρέπει να έχουμε εξασφάλιση οικονομική από τα κράτη-μέλη. Γιατί αμέσω αμέσως, αμέσως από τα 30 προγράμματα θα φτάσουμε στα 20 ή τα 10. Και αυτό θα είναι πιο πρακτικό να εφαρμοστεί. Χωρίς ε, οικονομικές συνέπειες όλοι θα θέλουν να συμβάλλουν στο πρόγραμμα αλλά κανένας δεν θα θέλει να πληρώσει. Αν θέλουμε λοιπόν να ενώσουμε την Ευρώπη, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα διέξοδα και πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα δύο, με τα διασυνοριακά συγγνώμη, ε, τμήματα των προγραμμάτων. Εμείς θέλουμε η Ευρώπη να ε, συνεργαστεί και σε αυτό θα πρέπει να επενδύσουμε και αυτό προς το παρόν δεν γίνεται. Γι' αυτό εδώ εγώ δεν λέω για περαιτέρω πηγές χρηματοδότησης. Τα ΣΔΙΤ ε, εντάξει, τα συζητάμε εδώ και 20 χρόνια και παρόλα αυτά τίποτα δεν έχει γίνει. Ε, ούτε για το διορθωτικό ταμείο θέλω να μιλήσω, ούτε για το, για το Ταμείο Συνοχή για την κινητοποίηση των διευρωπαϊκών ε, δικτύων. Απλώ πρέπει να δούμε αν έχουμε σωστή στοχοθέτηση. Ισπανία, α πούμε, ένα, ε, το αρνητικό ε, παράδειγμα από την Ισπανία είναι ότι από την, από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, χτίστη δημιουργήθηκαν, κατασκευάστηκαν ε, σιδηρόδρομοι εξαιρετικοί με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 80%. Αλλά αν πάρει κανείς το τρένο, κάθε βρίσκει συχνά πάρα πολλά ε, φορτηγά ε, γιατί υπάρχουν πολλοί παράλληλοι δρόμοι που κόβουν του σιδηροδρόμου, τέμνουν τι συνδρομικέ γραμμέ και κάθε τόσο σταματάει η κυκλοφορία για να περάσουν τα φορτηγά. Έχουμε εξαιρετικέ υποδομέ λοιπόν, τι έχουμε χρηματοδοτήσει, αλλά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Δηλαδή είναι ανόητο αυτό. Και ιδιωτικά κανένα δεν ήθελε να το κάνει. Κανένα δεν θα αγόραζε μια Mercedes, θα την έβαζε μπροστά στο σπίτι του και θα, θα μα έλεγε Δεν μπορώ να την κυκλοφορήσω, θα την κυκλοφορώ καλύτερα με το παλιό μου Fiat. Γερμανία. Από, Βερολίνο, από Βερολίνο προς Παλέρμο. Εξαιρετικοί οι δρόμοι, ε, περνάνε και μέσα από το, από το δάσος της ε, Έχουμε δώσει πάρα πολλά χρήματα για να γίνει αυτό, 15 χρόνια πήρε να γίνει, αλλά ο δρόμος από εκεί και μετά, από τα, όταν περνάμε, στα αυστριακά, περνάμε τα αυστριακά σύνορα, δεν υπάρχει ούτε μια γραμμή. Ή ε, Ρότερνταμ Γένοβα έγινε το τούνελ στην Ελβετία, το οποίο είναι έτοιμο. Και οι Γερμανοί δεν έχουν κάνει τους τους, ε, τις σιδηροδρομικές γραμμές, παρόλο που ήταν δεσμευμένοι να, και είχαν, προγραμματίσει να είναι έτοιμο. Όλα αυτά, καταλαβαίνετε, είναι τρελά. Νομίζω ότι με κάποιο τρόπο θα πρέπει να αποκλείουμε τις χώρες εάν δεν τηρούν τις, ε, ε, ε τις ε, συμβατικές τους υποχρεώσεις. Γι' αυτό συμφωνώ με αυτό που, που, που είπε ένα συνάδελφο πριν, ότι αν, οι, αν τα κράτη-μέλη δεν ε, τηρούν τι υποχρεώσει του, να του αφαιρεί τη χρηματοδότηση. Μόνο έτσι καταλαβαίνουν τα κράτη-μέλη. Λοιπόν, πρέπει να αποφύγουμε τα αδιέξοδα. Υπάρχουν πάρα πολλά ε, προγράμματα, πάρα πολλά κονδύλια. Μπορούμε να, να, να εξοικονομήσουμε χρήματα και δεν ξέρουμε ότι ας πούμε στο Αμβούργο υπάρχει πρόβλημα. Στοκχόλμη, Κοπενχάγη, από το Ρόστοκ προς Βερολίνο, Φραγκφούρτη, προς Βιέννη θα πήγαινε ο δρόμος, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να περάσει από το, από το Αμβούργο και θέλουμε εμείς να λύσουμε το πρόβλημα βάζοντας ακόμη περισσότερη κυκλοφορία να περνάει από το Αμβούργο που ούτως ή άλλως είναι μποτιλιαρισμένο. Κανένα δεν μπορεί να πληρώσει όλα αυτά τα ιδέατα ε, προγράμματα που φανταζόμαστε. Γιατί συνέχεια λέμε θέλουμε περισσότερα λεφτά, θέλουμε περισσότερα λεφτά. Αν δεν δούμε ποιε ήταν οι συνέπειε από αυτό που πήγε στραβά, δεν θα βρούμε πρόβλημα, δεν θα βρούμε λύση. Δεν θέλουμε περισσότερα χρήματα, θέλουμε περισσότερη εξυπνάδα. Ε, Εντάξει, όλα τα προγράμματα είναι σημαντικά, αλλά πρέπει να σκεφτούμε τι έχουμε κάνει λάθος και να μάθουμε από τα λάθη μας. Δεν μπορούμε συνέχεια να ευχόμαστε να αυξηθούν τα κονδύλια. Ευχαριστώ. Και eh, Ο κύριος Ζήλα, ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ είμαι πολύ ευτυχής που καλωσορίζω εκπροσώπου τη Επιτροπή ΣΟΥΡ, την πρόεδρο, καθώς και τον εισηγητή Εργάζομαι στην Επιτροπή Crisis. Ε, Και να μην κάνετε εσεί το ίδιο λάθο που κάναμε εμεί στη δική μα ειδική επιτροπή στην αρχή. Ξεκινήσαμε από διάφορα έγγραφα εργασίας, μικρά, σύντομα, αλλά η έκθεση απέτησε από τους συναδέλφους να στείλουν 1.700 τροπολογίες. 90% από τις τροπολογίες απερίφθησαν πριν τις ψηφοφορίες. Οπότε καταφέραμε να μειώσουμε τον αριθμό των τροπολογιών που πήγαν για ψηφοφορία στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια. Τώρα πηγαίνοντας πίσω στις δικές σας εργασίες, πολύ δύσκολο το έργο σας, πάρα πολύ δύσκολο. Δύσκολο να εξηγήσει κανείς τους φορολογούμενους γιατί οι δημοσιονομικές προπτικές ε, πρέπει να έχουν πολύ μεγάλα ποσά μετά το 2014. Πολλές κυβερνήσεις ξεκίνησαν με προγράμματα λιτότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα κράτη-μέλη και είναι πολύ δύσκολο να πείσει κανεί το λαό ότι χρειαζόμαστε χρήματα για τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεω, ξεκινώντας ήδη από το 2011 μέχρι το 2014. Διότι η κοινωνία είναι πολύ απεσιόδοξη. Σε αυτή τη φάση μάλιστα. Όσον αφορά την γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών, αυτήν που ετοιμάζουμε, Είμαι κάπως διχασμένος. Από τη μία πιστεύω ότι η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία θα πρέπει να ενισχυθεί και να υπογραμμιστεί. Απ' την άλλη όμως, αυτή η προστιθέμενη αξία πάντα θα είναι υψηλότερη στη Δυτική Ευρώπη, όπου είναι πιο πυκνοκατοικημένη, όπως είναι η Γερμανία, η Γαλλία, η περιοχή των Άλπαιων, όπου εκεί πάντα θα έχουμε μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία όσον αφορά τη δημιουργία μεταφορικών δικτύων εν συγκρίση με περιφερειακές ζώνες. Και τα νέα κράτη-μέλη, είναι λάθος διατύπωση, συμφωνώ, λάθος έκφραση. Γιατί? Διότι τα νέα κράτη-μέλη έχουν πολύ αδύναμες ε, μεταφορικές υποδομές παραδοσιακά συνδεόταν με το παλιό κομμουνιστικό μεταφορικό δίκτυο. Οπότε γεωγραφικά και τεχνολογικά είναι πίσω. Δύσκολο να διασυνδεθούν με την Δυτική Ευρωπαϊκή Ένωση και χρειαζόμαστε αυτές τις διασυνδέσεις. Η προστεθέμενη αξία μας πάντα θα είναι χαμηλότερη και η επιστροφή των χρημάτων των επενδύσεων θα είναι χαμηλότερη στην Ανατολική Ευρώπη από τη στη Δυτική. Τι πρέπει να κάνουμε. Στο σημείο 9 της γνωμοδοτήσεως ζητάμε συγκεκριμένη ποσά για προγράμματα TNT για τα νέα κράτη-μέλη. Συμφωνώ με αυτό, όμως ε, γνωρίζουμε ότι η δημοσιονομική πόροι των κυβερνήσεων είναι άκρως περιορισμένοι. Στις βαλτικές χώρες υπάρχει μόνο ένα πρόγραμμα TNT το, για σιδεοδρόμου, το Rail Baltic, αν θέλουν οι κυβερνήσεις χρηματοδοτήσουν το πρόγραμμα, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να πάρουν χρήματα από άλλου τομεί πολιτική, όπως είναι η γεωργία ή άλλοι σημαντικοί οικονομικοί τομείς. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο εγώ να το υποστηρίξω αυτό το σημείο. Οι πολιτικοί μας ε, περνάνε δύσκολες ώρες. Ε, αναφερόμενοι τώρα στις μεταφορές, πρέπει να πούμε ότι υπήρξαν διασυνδέσεις στη χώρα, στις βαλτικές χώρες με το ρωσικό σύστημα. Και είναι δύσκολες οι επαφές με τους Ρώσους εταίρους μας. Αυτοί πιστεύουν ότι επενδύσεις για τη Rail Baltica δεν χρειάζονται. Ότι το σύστημα των βαλτικών χωρών, το σιδηροδρομικό, δεν χρειάζεται να συνδεθεί με τη Δυτική Ευρώπη, διότι έχουμε σημαντικές εμπορικές σχέσεις με τους Ρώσους ακόμα. Οπότε οι συνδρομικές μας διασυνδέσει είναι κυρίως μεταξύ βαλτικών χωρών και Ρωσίας. Από Δυσμάς προς Ανατολάς. Και όχι από εμά προς Βορρά ή προς Νότο. Αλλά είναι σημαντική αυτή η διασύνδεση για μας με τα συνδρομικά συστήματα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Είναι περιπλοκότατα ζητήματα και θα προσπαθήσω να συμβάλλω λίγο σε εργασία επιτροπής. Σύρ, ο κύριος Ρίκε έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς ε, να ευχαριστήσω τη Γιούτα και το Σαλβαδόρ για την παρουσία τους και για τη δουλειά που κάνουν. Έχω ένα σχόλιο γενικό. Η Επιτροπή Μεταφορών εργάστηκε όσον αφορά τη διοργάνωση των μεταφορών στην Ευρώπη, ετοίμασε οδηγίες ή κανονισμούς που επιτρέπουν το άνοιγμα της αγοράς, τη λειτουργικότητα, χρήση των δικτύων κάναμε ό,τι μπορούμε για να λειτουργεί το μεταφορικό σύστημα. Αλλά θα πρέπει το μεταφορικό σύστημα να υφίσταται. Δηλαδή να υπάρχουν υποδομέ και να είναι προσαρμοσμένε σε όλη την επικράτεια τη ενώσεω. Κάτι που ανέφερε εξάλλου ο συνάδελφο. Και, και τις ανατολικές χώρες, πιο ανατολικέ, δεν θα πω νέα κράτη-μέλη. Και εκεί πρέπει να λειτουργήσει το σύστημα. Η Επιτροπή Μεταφορών λοιπόν είναι παρούσα μαζί με τον τουρισμό έχει σημαντικό ποσοστό του ΑΕΠ, πολλά διακυβεύονται και στον τομέα του περιβάλλοντος. Αυτή η Επιτροπή λοιπόν δεν έχει τη δυνατότητα την επιχειρησιακή, τη λειτουργική όσον αφορά τις επενδύσεις που χρειάζονται για τον τουρισμό, ε, για το, τις μεταφορές. Έχουμε περίπου ένα δισεκατομμύριο, τώρα άντε 900 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο έχουμε όσον αφορά την εκτελεστική υπηρεσία του, των δικτύων και τα διακευόμενα όσον αυτο το σχεδιασμό φτάνουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Άρα πρέπει να στραφούμε αλλού για να βρούμε χρήματα για τις μεταφορικές υποδομές. Υπόθηκε κάτι επίκαιρο. Επιτροπή ρεζί θα πρέπει να βρει τα περισσότερα μέσα για να μπορεί να τα διαθέσει στις μεταφορές. Και το λέω διπλωματικά, διότι οι συνάδελφοι της, Επιτροπής, ε, της Περιφερειακής Επιτροπής δεν θέλουν να χάσουν πιστώσεις και έχουν συγκεκριμένο όραμα. 28% των πιστώσεών τους πηγαίνουν για υποδομές με προστιθέμενη αξία ευρωπαϊκή με συμπερίφθη στα δίκτυα, αλλά κατά τα λοιπά πηγαίνουν αλλού. Η βάση της περιφερειακής πολιτικής ε, δεν είναι ειδικά οι διασυνδέσεις σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Ζητάμε από τους συναδέλφους Επιτροπής Ρέζη να αλλάξουν κάπως την οπτική τους γωνία και πώς λειτουργούν όσον αφορά τη διάθεση πόρων. Δεν θα τους πάρουμε τις πιστώσεις, αλλά θέλουμε να συζητήσουμε μαζί τους. Ε, δεύτερη ενδεχόμενη πηγή πόρων είναι οι νέοι πόροι. Κάτι που συζητούν πολύ στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Δεν πρέπει να ειδωθούν αυτά σαν νέοι φόροι απαραίτητα. Νέες, νέες πηγές για χρηματοδότηση υποδομών. Ευρωβινιέτα, παραδείγματο χάρη. Είναι προχωρημένη αυτή η ιδέα. και δεν επηρεάζονται σε μεγάλη κλίμακα ειδικέ μεταφορέ από τον πόρο. Αλλά έχουμε δεύτερη ενδεχόμενη πηγή χρηματοδοτήσεω. Δεν μπορούμε να το συζητήσουμε όμω άμεσα αυτό. Τρίτον, υπάρχουν πηγές νέε που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προπολογισμού για του σκοπούς μας. Το λέω απευθυνόμενο προς συναδέλφου τη Επιτροπή Προπολογισμών άνευ σχολείου Γιούτα από ό,τι βλέπω. Υπάρχουν περιορισμοί με τη συνθήκη της Λισαβόνας, υπάρχουν όμως νέες ευθύνες και σε αυτό το πλαίσιο δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στις νέες ευθύνες. Άρα δεν είναι εύκολη αυτή η αναδίπλωση. Έχουμε πρόβλημα αν υπάρχουν πόροι και δεν μπορούμε να του ελέγξουμε, απ' έξω είναι δύσκολο να βρούμε νέου πόρου και οι, ανα... οι μεταφορές κονδυλίων, οι αναδιπλώσει κλπ. Οι είναι κάτι πολύ δύσκολο. Για τον τουρισμό τώρα. Υπερασπίστηκα στις προτάσεις όσο μπορούσα. Μετά τη συνθήκη της έχουμε νέα αρμοδιότητα του τουρισμού. Σημαντικό ποσοστό, σημαντικός τομέας για την οικονομία, για απασχόληση και ΑΕΠ. Μπορούμε έτσι με τριοπαθώς δειλά-δειλά να εισαγάγουμε κάποια προγράμματα πιλωτικά. διότι όπως υπενθύμησε και ο Σαλβαδόρ, δεν υπάρχει συμφωνία με το Συμβούλιο όσον αφορά τη χρηματοδότηση των νέων ευθυνών που απορρέουν τις συνθήκε τη Αβώνα. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία προοπτική όσον αφορά τον προπολογισμό για τον τουρισμό πριν το 2013. Τα ίδια θα συμβούν και το 12 και το 2013. Και η μόνη δυνατότητα που έχουμε όσον αφορά το σημαντικότατο θέμα αυτό είναι στα πλαίσια των δημοσιονομικών προπτικών 2014-2021 να πείσουμε την Επιτροπή Προλογισμών και κυρίως τα κράτη πείσουμε ότι δεν αξίζει τον κόπο να δίνει κανείς ευρωπαϊκές ευθύνες νέες χωρίς να διατίθενται και αναγκαίοι πόροι. έχει 20% του ΑΕΠ, 35% ε, της ρήπανση στον τομέα μας με αυτό που ασχολούμεθα και δεν λειτουργεί καλά τομέα. Σε ευρωπαϊκή κλίμακα χρειάζονται μέτρα. Είναι στατική σημασία η Επιτροπή για τις υποδομές και δεν έχει χρήματα. Και αυτό είναι πάρα πολύ παράξενο. Η κυρία Τσικάου έχει το λόγο. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ και την κυρία Χάουκ και τον κύριο Γκαρίδα Πογέδο και θα ήθελα να ζητήσω στην ε, έκθεση αλλά και στην εφαρμογή της ε, έκθεσης να υποστηρίξετε την ε, Επιτροπή μας ώστε ένα σημαντικό τμήμα του ευρωπαϊκού προπολογισμού να αποδοθεί στον, στις μεταφορές, στον τομέα των μεταφορών. Είναι σημαντικό και για την ανταγωνιστικότητα αλλά και για την ε, κοινωνική ανάπτυξη της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης στην Επιτροπή Τραν εδώ ε, λυπούμεθα που η Κομισιόν μέχρι τώρα δεν έχει δημοσιεύσει τη Λευκή Βίβλο για τις μεταφορές. Επίσης, ε, λυπούμεθα για τις διαπραγματεύσεις ε, για τον ε, επόμενο προπολογισμό, οι οποίες ξεκίνησαν και για το ε, μέλλον της ε, πολιτικής της, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Και επίσης δεν έχουν ληφθεί υπόψη α, κάποια προγράμματα, τα TNT, το Μαρκοπόλο, το τον ΑΙΑΔΕΣ. Ούτως ή όλος η περίοδος των δημοσιονομικών προοπτικών ολοκληρώνεται. Αλλά θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και μετά το 2013, όπου λύγει η περίοδος αυτή. Είναι σημαντικό να έχουμε έναν κατάλογο όλων των, δημοσιο... όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων που έχουμε στη διάθεσή μας για να δούμε τι χρηματοδοτείται ή τι θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί στον τομέα των μεταφορών και από πού. Για το Γαλιλαίο τώρα είναι στρατηγική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να υπάρξουν ε, χρηματοδοτικοί πόροι για αυτό. Σκέφτομαι εδώ τη χρηματοδότηση ε, ερευνητικών Ινστιτούτων που σχετίζονται με αυτό για την τεχνολογική, τεχνολογική ανάπτυξη δεν αντικατοπτρίζεται στον ε, προπολογισμό. Η αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών επίσης, σε σχέση και με τις μεταφορές. Ούτε γι' αυτό βλέπουμε κάποια γραμμή του προπολογισμού. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να σας ρωτήσω η έκθεσή σας δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει και μια απάντηση για το ερώτημα πώς τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια για τις μεταφορές. Ποιες συστάσεις θα πρέπει να κάνουμε στην Κομισιόν έτσι ώστε στην εφαρμογή του επόμενου προϋπολογισμού να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα αυτού του ταμείου. Και μια τελευταία παρατήρηση για το TEN-T υπάρχει συγχρηματοδότηση. Αν τώρα μιλούμε για το μέλλον των διευρωπαϊκών δικτύων, των TEN-T, η Κομισιόν αναφέρει και τους εθνικούς προπολογισμούς. Νομίζω ότι σημαντικό θα ήταν να εξασφαλίσουμε ότι η συγχρηματοδότηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων θα αντικατοπτρίζεται και στους εθνικούς προπολογισμούς. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στους ομιλητές για να απαντήσουν, ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης MOVE έχει έρθει και έχει ακούσει τη συζήτησή μας. Θα ήθελε λοιπόν να παρέμβει. Ε, ε, ευχαριστώ πολύ, Μπράιαν. Ευχαριστώ την κυρία Χάου και τον κύριο Γκαρίγα για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Προφανώς δεν είμαι εδώ για να σας αποκαλύψω το τι θα θέσει επιτάπητος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τον προϋπολογισμό. Θέλω να πω όμως μερικά λόγια σχετικά με το θέμα. Το θέμα μας, το χαρτοφυλάκιό μας, τις μεταφορές. Να υπενθυμίσω τρία στοιχεία. Ήδη τα θύμισες, Μπράιαν. 45% ΑΕΠ 14% δαπανών νοικοκυριών πάνε στις μεταφορές και αυτό είναι τμήμα του τουρισμού και κάτι άλλο που θα πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι η Ευρώπη ηγείται σε παγκόσμια κλίμακα στον τομέα των μεταφορών. Επιμελητή, οργάνωση. Θαλάσσιες μεταφορές. 40% των παγκοσμίων στόλων, του παγκόσμιου στόλου είναι ανήκει σε Ευρωπαίους αερομεταφορές, τρένα εμψηλής ταχύτητας, διαχείριση, συστήματα διαχείριση της κυκλοφορίας κλπ. Υγούμεθα στον κόσμο και κινδυνεύουμε να χάσουμε τη θέση μας αυτή, διότι όπως είπατε κάποιοι, άλλες περιοχές του κόσμου, Κίνα, είπα σπρώχνουν πολλές επενδύσεις στις μεταφορές είναι κρίσιμη, είναι κομβικό σημείο αυτό. Διότι όπως αναφέρθηκε πρέπει να ετοιμάσουμε ριζικές αλλαγές του μεταφορικού συστήματος διότι φεύγουμε το πετρέλαιο, απομακρυνόμαστε. Είτε για λόγους κλιματικούς ή γιατί, γιατί σπανίζει το πετρέλαιο ή θα γίνει πολύ ακριβό, πρέπει να αλλάξουμε όσον αφορά την αντιμετώπιση των μεταφορών. Τώρα είναι η ώρα όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει πραγματικά ευρω... προγράμματα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, διότι θα γίνουν αλλαγές. Γι' αυτό ε, σκεφτόμαστε τα διευρωπαϊκά δίκτυα και τα βλέπουμε με διαφορετικό μάτι. Θέλουμε να δημιουργήσουμε βασικό δίκτυο που ξέρετε με διόδους, διαδρόμους που συνδέεται με κομβικά σημεία, σημεία εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, διαδρόμους ε, διαμεταφορικούς, με διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς, ευφυείς μεταφορές, θέλουμε πράσινες μεταφορές, ενταξιακές μεταφορές, όλες οι πτυχές οι βιώσιμες θέλουμε, οι πτυχές να μπουν στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Ακούσαμε πολλά να λέγονται για την Επιτροπή Μεταφορών, την Περιφερειακή Επιτροπή. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινόμαστε προς σφαιρική, ενιαία αντιμετώπιση. Συνεργαζόμαστε με τους συναδέλφους για τα περιφερειακά θέματα. Θέλουμε κοινό πλαίσιο οικονομικό. 43 δις από τη συνοχή και τα περιφερειακά ταμεία πάνε στις μεταφορές. 8 δισεκατομμύρια από τα διευρωπαϊκά δίκτυα. 60 δις κινητοποιούμε μέσω ε, χορηγήσεων, μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, τη μορφή δανείων. 200 δισεκατομμύρια χρειαζόμαστε για τα δίκτυα συνολικά. Αρκετά χρήματα. Κινούμαστε μαζί. Και στο μέλλον θα υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη συνεργασία. να απομακρυνθούμε από το μύθο ότι τα διευρωπαϊκά δίκτυα αφορούν ε, κάτι αφηρημένο. Δεν θα υπήρχε ο Γαλιλαίος αν δεν υπήρχε το, υπήρχαν τα ευρωπαϊκά δίκτυα. Πιλωτικό πρόγραμμα 15. Πρώτα δώσαμε χρήματα για την έρευνα και μετά διευρωπαϊκά, με πόρους για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Διαχείριση σιδηροδρομικών συστημάτων χρησιμοποιούνται σε όλο τον κόσμο. Χιλιάδε χιλιόμετρα ευρωπαϊκή τεχνολογία χρησιμοποιούνται εκτό Ευρωπαϊκή Ενώσεω. 6 με 7 χιλιάδες και το 2020 ελπίζουμε 30 χιλιάδες. Έρευνα, καινοτομία, μπήκαν σε αυτό, επιδείξεις και χρήματα διευρωπαϊκών δικτύων για την εγκατάσταση. Συστήματα ενημέρωσης, ε, συστήματα ασφάλειας. Ε, μπαίνει πολλή προσπάθεια, πολλά ευφυή e συστήματα στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Και πολλοί νους και σκέψη. Καινοτομία. Αναφέρθηκα τι πρέπει να κάνουμε. Χρειαζόμαστε εναλλακτικά καύσιμα, καθαρότερα οχήματα, εναλλακτικές υποδομές δηλαδή προγράμματα καινοτομία και έρευνα. Θα εστιαστούμε βασικά σε αυτά, πιστεύω, τα βασικά θέματα. Και μετά καινοτόμο χρηματοδότηση, γιατί θα λείπουν τα χρήματα. Θέλουμε καινοτόμε μεθόδου χρηματοδοτήσεω. Ένα από τα καλά παραδείγματα, ελπίζουμε, θα είναι ένα, να έχουμε κάποιο ομόλογο ε, για τα προγράμματα και ίσω στι μεταφορέ θα εγγυηθούμε σε αυτό το τομέα και για να δουλέψουν αυτά που θέλουμε ε, στα πλαίσια του προγράμματος ΣΕΖΑΡ. 2 δισεκατομμύρια ευρώ κινητοποιήθηκαν, 600.000 από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το προβλησμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, 600-700 από το Eurocontrol και το τελευταίο τρίτο από το τομέα. Υγηθήκαμε και εκεί όσον αφορά τα εναλλακτικά προγράμματα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε που μου δώσατε τη δυνατότητα να σχολιάσω κάπως τα όσα υπόθηκαν. Ευχαριστώ κύριε Ρόιτα. Ποιος έχει σειρά, ο Σαλβαδόρ. Θες να συνοψίσεις. Ο Πρόεδρος. Όταν έχεις αμφιβολίες ρώτα τον Πρόεδρο. Ευχαριστώ. Ήρθαμε σήμερα για να ακούσουμε αυτά ακριβώ Αυτά που λένε οι συνάδελφοι αυτά που λέει ο Γενικός Διευθυντής. Θα ήθελα να σχολιάσω λίγο ποια είναι η εντολή που έχει η Επιτροπή μας, η Επιτροπή ΣΥΟΡ. Έχουμε μια τελείως διαφορετική ε, εντολή εμείς από την Επιτροπή Crisis. Ε, ε, έχουμε δηλαδή ένα στόχο, τον Ιούνιο του 2011, αυτή την έκθεση να την πάμε στην Ολομέλεια. Και ελπίζουμε να την ψηφίσουμε και με μεγάλη πλειοψηφία και η Επιτροπή μας μετά θα έχει ολοκληρώσει το έργο της. Δεν θα ζητήσουμε παράταση. Έχουμε τόσο λίγο χρόνο για ένα τόσο τεράστιο θέμα, αναφυσβήτητα, που δεν ασχολούμαστε καθόλου με κάποιες άλλες ε, μικρότερες εκθέσεις, λίγο πιο πριν, λίγο πιο μετά. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που η, Ευρωπα... η, η θέση του Κοινοβουλίου περιγράφεται για τις, υπόλοιπες, για τις ε, μελλοντικές δημοσιονομικές προοπτικές πριν υποβάλει η Κομισιόν την πρότασή της. Αυτή την ε, δυνατότητα την είχαμε λόγω του ότι ε, συνέβαλαν διάφορα πράγματα, ξεκίνησε αργά η Κομισιόν τη δουλειά τη και άλλοι παράγοντες, αλλά χρησιμοποιήσαμε εμείς την ευκαιρία που μας δόθηκε και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να την αξιοποιήσουμε με ένα καλό αποτέλεσμα στο τέλος των Ιούνιου του 2011. Αυτό που κατάλαβα καλά είναι για τον τομέα της, ε, των μεταφορών ότι ισχύει ότι έχουμε μεγάλη προσθέμενη αξία, ότι θέλουμε να υπάρξει ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς με έναν ορθώς λειτουργώντα τομέα, ε, λειτουργούντα τομέα μεταφορών, ότι πρέπει επιγόντως να απαλείψουμε τα διέξοδα και πρέπει να, να δώσουμε βαρύτητα στις διασυνοριακές συνδέσεις. Ή να τις, να ενισχύσουμε, να τις βελτιώσουμε εκεί που υπάρχουν αλλά δεν λειτουργούν πολύ σωστά. Αυτό που είναι επίσης σαφές και προέκυψε και από αυτά που είπε ο Γενικός Διευθυντής, είναι ότι αν αν προωθήσουμε τη στρατηγική 2020, έχουμε, πρέπει να προωθήσουμε και τους, και τους τρεις ε, στόχους. Πρέπει να τους βλέπουμε όλους από κοινού. Δεν μπορούμε να λέμε ε, θα πάρουμε μόνο, ξέρω εγώ, την ανταγωνιστικότητα και αυτό θα είναι ο στόχος μας να την αυξήσουμε, να την βελτιώσουμε και η, τα προβλήματα της, ε, των μεταφορών μετά. Πρέπει να τα δούμε ταυτόχρονα και τη βιωσιμότητα και την κοινωνική συμπερίληψη. Όλα πρέπει να τα, να τα σκεφτόμαστε από κοινού. Από μόνα, του δεν μπορούν να λυθούν τα, από τα προβλήματα. Πρέπει να τα, δούμε όλα μαζί. Και σωστά το λέει και η Κομισιόν και οι πολιτικές επίσης πρέπει να έχουν κάποιες κοινέ κατευθυντέρε γραμμές. Δεν μιλούμε μόνο για, τη, για τα περιφέρεια και για, την, για τις μεταφορές, μιλούμε και για τη γεωργική πολιτική, για την αναπτυξή του υπαίθρου, και για αυτά χρειάζεται μια κοινή πολιτική και για την ανάπτυξη πέθρου χρειάζονται μεταφορές. Όλα αυτά λοιπόν διασυνδέονται. Να σκεφτούμε ας πούμε τις έξυπνες πόλεις. Για να έχουμε έξυπνες πόλεις χρειαζόμαστε έξυπνες μεταφορές. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα έχουμε συνεχώς υπόψη μας. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε το ένα υπέρ του άλλου. Το θέμα της αιρεσιμότητας που ετέθη. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αλλά δεν μπορούμε να το δούμε μόνο μέσω του προπολογισμού. Θα έχουμε με την έκθεση του Σαλβαδόρ ε, μια δομή έτσι για τον προπολογισμό, για το πώς θα είναι δηλαδή οι ε, δημοσιονομικές προοπτικές και πώς θα έχουν οι πολιτικές και ποιο τμήμα θα αποδοθεί πού από τον ε, προπολογισμό. Αλλά μετά, όταν θα έχουμε τα προγράμματα και, τα, και τα σχετικές δαπάνες θα πρέπει να τα ξανασυζητήσουμε. Να δούμε δηλαδή υπό ποιε προϋποθέσεις και ποιους όρους θα πρέπει να θέσουμε. Η Κομισιόν στην έκθεσή της μιλά για τη λειτουργία των υπαρχουσών ε, δημοσιονομικών προπτικών. Πρέπει όμω να δούμε και τι επόμενε δημοσιονομικέ προοπτικέ και να δούμε ποια είναι τα λάθη που κάναμε σε τούτε για να μάθουμε από τα λάθη μα. Και έρχεται η Κομισιόν και καταλήξει στο συμπέρασμα ότι σε κάθε τομέα πολιτικής που ε, συνδέεται με, ε, ε με επιδοτήσεις θα πρέπει να, συν, να συναυθούν ε, συμβάσεις με, την, ε, με τα κρατημέλη, με, τα συμβαλόμενα μέρη, όπως κάνουμε στα ΣΔΙΤ, κάπως έτσι και ταυτόχρονα, δεν το λέει βέβαια η Κομισιόν, το λέω εγώ και θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, πρέπει να ε, προβλέψουμε και κυρώσεις για καταπατήσεις. Δεν μπορούμε δηλαδή να έχουμε συμβάσεις χωρίς να ξέρουμε τι γίνεται αν δεν τηρηθούν οι συμβάσεις. Γιατί αλλιώς είναι ε, επιφανειακές, είναι άχρηστες οι συμβάσεις αυτές. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν και κυρώσει, πρέπει να υπάρχουν πρόστιμα, πρέπει να υπάρχει κάποια ποινή. Φυσικά όλοι θέλουμε να έχουμε μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία από αυτό το 1% του ΑΕΠ που μας αναλογεί. Όσο περισσότερη προστιθέμενη αξία μπορούμε να στραγγίξουμε από αυτό το 1%, αυτό θα κάνουμε. Σημειώσαμε λοιπόν όλα σας τα σχόλια και θα τα έχουμε υπόψη μας. Τελεία. Michael, Michael always likes to have the last word. Πάντα ο Μάικλ θέλει να λέει την τελευταία κουβέντα. Εκ μέρου τη Επιτροπής ευχαριστώ τη Γιούτα και το Σαλβαδόρ. Σας ευχαριστώ που ήρθατε και διαθέσατε χρόνο. Ακούσατε τα μέλη, τι απόψει του και προσβλέπουμε σε συνεργασία μαζί σας μαζί σας του χρόνου προθεσμία για υποβολή τροπολογιών για το σχέδιο γνωμοδοτήσεώς μου είναι 8 Δεκεμβρίου. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή Μεταφορών τον Ιανουάριο για να υποβάλουμε τη γνωμοδότηση στους φίλους μας στη Νομική Επιτροπή ταχύτερο δυνατό, στη ΣΟΥΡ μάλλον, συγγνώμη, ταχύτερο δυνατόν. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και μη λησμονείτε, λέει η κυρία Χάουγκ, ότι τον Φεβρουάριο είναι, θα συζητήσει για τα TNT η Επιτροπή. Λοιπόν, σας προσκαλούμε εκεί, θα συζητήσει η Επιτροπή μας τα TNT για μια ακόμη φορά. Okay, colleagues, we've now got to... Συνάδελφοι, πρέπει να συζητήσουμε το θέμα της ε, συμφωνίας με την Βραζιλία για τις αρωματοφόρες αεροπορικές μεταφορές. Η κυρία Τσικάου λοιπόν έχει το λόγο. Για τις αεροπορικές μεταφορές. Uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόκειται για σημαντική συμφωνία. We'll move them out. We'll keep going. Uh, uh, Έχουμε να κάνουμε με μια διεθνή πολύ σημαντική συμφωνία για την πολιτική αεροπορία. Πρόκειται για συμφωνία που υπεγράφει μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βραζιλίας. Πρέπει να αναφέρω κάποιους αριθμούς για τους συναδέλφους. Η Βραζιλία είναι πάρα πολύ σημαντική για την Λατινική Αμερική. Είναι η Ευρώπη ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίως ο μεγαλύτερος επενδυτής στη Βραζιλία είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν αναφερθούμε στις επιπτώσεις αυτής της συμφωνίας για τον τουρισμό, μπορούμε να αναφέρουμε το γεγονός ότι για ε, Practic, numărul acesta reprezintă 35% για ένα εκατομμύριο και ε, επιβατών ε, τουριστών από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς, το, προς τη Βραζιλία μιλούμε για ένα 35%. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 22% των διεθνών πτήσεων. Είναι λοιπόν ο πλέον σημαντικός ή ο δεύτερος πλέον, σημαντικός, πλέον σημαντική αγορά προς την Αργεντινή. Και στην τρίτη θέση είναι η ΙΠΑ. Επίσης η Βραζιλία είναι στη δεύτερη θέση στον κόσμο για τον, στον, σε ό,τι αφορά τον αριθμό των αεροδρομίων μετά τις Ηνωμένε Πολιτείες με περίπου 15.000 αεροδρόμια. Και μετά 15.000 αεροδρόμια έχει, έχουν η και 4.000 αεροδρόμια έχει η Βραζιλία. Επίσης, οι θετικές συνέπειες της συμφωνίας στον τουρισμό είναι σαφής επειδή ακριβώς υπάρχει και μια απελευθερωμένη αγορά που επιτρέπει την ε, ελεύθερη ε, διακίνηση των ε, πτήσεων μεταξύ Ευρώπης και Βραζιλίας. 145 εκατομμύρια, από τα οποία 86 εκατομμύρια είναι κέρδος από τον τομέα του τουρισμού στην ε, Βραζιλία και 49 είναι το κέρδος για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές οι συνέπειες ε, αντικαθιστούν κάποιες ρήτρε οι οποίες υπάρχουν ήδη σε 15 διμερείς συμφωνίες. Υπάρχουν 15 διμερείς συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βραζιλίας προς το παρόν. Αλλά επειδή υπάρχει και μία απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μόνη υπεύθυνη για, την, για τις μεταφορές. Οπότε οι συμφωνίες τώρα ρυθμίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω μια συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βραζιλίας. Αυτές οι ρήτρες αφορούν τον ορισμό ενός, μιας εταιρείας η οποία είναι εγκεκριμένη και που μπορεί να δραστηριοποιείται στον εναέριο χώρο της Βραζιλίας. Είναι σημαντικό αυτό και για την ασφάλεια και, για το, και το άρθρο 4 αφορά ε, την, φορολογία των ε, καυσίμων των αεροπλάνων. Επίσης, ένα άλλο που είναι πολύ σημαντικό είναι η εναρμόνιση με, τους, με τα πρότυπα ανταγωνισμού έτσι ώστε όλες οι εταιρείες αεροπορικών μεταφορών από την Ευρώπη να έχουν ίδια πρόσβαση στην, στη βραζιλιάνικη αγορά. Είναι επίσης σημαντικό οι διμερείς, σχε... οι διμερείς συμφωνίες να εφαρμόζονται. Η συμφωνία που έχουμε και συζητούμε σήμερα δεν αντικαθιστά τις διμερείς συμφωνίες. Αυτό είναι σημαντικό. Αντικαθιστά μόνο κάποιες ρήτρε από τις διμερείς ε, συμφωνίες. Έτσι, ώστε να υπάρχει η μία ίση πρόσβαση χωρίς καμία διάκριση στην ε, αγορά των ε, αεροπορικών μεταφορών. Και κλείνοντας να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύεται και θα υπογράψει μία συμφωνία για τις αεροπορικές μεταφορές με την Βραζιλία και αυτή η συμφωνία είναι επίσης πολύ σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σταματήσω εδώ και θα προτείνω στους ε, συναδέλφους να υπερψηφίσουν την έκθεση αυτή έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε την ε, σύμφωνη γνώμη μας για την σημαντική αυτή συμφωνία. Βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας για σχόλια, ερωτήσεις κτλ. Ευχαριστώ πολύ. Να επενθυμίσω ότι είναι διαδικασία συμφώνου γνώμης αυτής. Δεν μπορούμε να τροποποιήσουμε το κείμενο της συμφωνίας μπορούμε να τροποποιήσουμε το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος ή να απορρίψουμε τη συμφωνία, αλλά δεν μπορούμε να το αγγίξουμε το κείμενο. Έτσι εξοικονομούμε και πολύ χρόνο. Να μην συζητάμε πράγματα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριος Τεσέρα. Αρχίζοντας θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Τσικάου, την εισηγητριά μας, για την έκθεσή της. Και αν με επιτρέπετε θα ήθελα να κάνω μόνο κάποιες πολύ σύντομες παρατηρήσεις για το θέμα αυτό και να πω πόσο σημαντικό είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να πω κάτι θεσμικού περιεχομένου. Χαιρετίζω την ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο θέμα αυτό για την έγκριση δηλαδή διεθνών συμφωνιών και κυρίως για θέματα τα οποία αφορούν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και συγκεκριμένα εδώ σε νέες μεταφορές, αλλά πρέπει να πω ότι λυπούμε και καταγράφω το γεγονός ότι ζητείτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πει την άποψή του αργά, αφού έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις. Άρα είναι πολύ περιορισμένος ο ρόλος μας. Επίσης ήθελα να πω ότι αυτή η οριζόντια συμφωνία την πολιτική αεροπορία είναι ένα μεγάλο άνοιγμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα δημιουργήσει ένα σύγχρονο πλαίσιο σχέσεων μεταξύ Βραζιλίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι λοιπόν πρωταρχή σημασία η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση να έχει και εδώ μία πολιτική συνεκτική δεδομένου ότι έχουμε να κάνουμε με τρίτη χώρα με την οποία θέλουμε να έχουμε συνεκτική πολιτική, πιο ανταγωνιστική, με ενιαία εσωτερική αγορά και να μπορεί να λειτουργεί με υγιείς κανόνες της αγοράς η Ευρώπη. Είναι σημαντικό. Επίσης θα πρέπει να επενθυμίζω ότι ο στόχος της μη διάκρισης και η τήρηση του δικαιώματος να έχουν κάπου την έδρα τους διάφορες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πρέπει να συνάδει με το υπάρχον σύστημα. Άρα γι' αυτό θα χρειάζεται να έχουμε μία σύγχρονη και ανανεωμένη αν θέλετε νομική βάση. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με, τώρα με ένα πρώτο βήμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα πρώτο βήμα μία σειρά βημάτων που θα πρέπει να γίνουν ε, και όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν με προοδευτικό τρόπο. Θα πρέπει να επικαιροποιήσουμε τις ε, συμφωνίες, τις διμερείς συμφωνίες όλες να τις αντικαταστήσουμε με κοινοτική συμφωνία και να μπορέσει στα πλαίσια αυτής της εργασίας η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να έχει όχι μόνο οικονομικά ωφέλη αλλά να συνάψει και στρατηγικής ε, σημασίας εταιρικές σχέσεις. Είναι επίση πολύ σημαντικό, εκτό από αυτή τη συμφωνία, να πούμε ότι έχει και οικονομικά ωφέλη αυτή η συνωνία. Ε, πλέον εκτίμακτα δεδομένου ότι θα είναι ποφελής για τους πελάτες, θα υπάρχουν φτηνότερα ειστήρια αν θέλετε για τους επιβάτες, ε, πιο ανταγωνιστικές τιμές και δεδομένου ότι έχουμε να κάνουμε με οικονομίες, μιλάμε για 300 με 400 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για τους, ε, οικονομίες για τους επιβάτες. Και βεβαίω θα έχουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο πολύ πιο ανοιχτό. Για αυτούς όλους τους λόγους και για τους λόγους που ανέφερε και η συνάδελφος κυρία Τικάου και εγώ κάνω έκκληση για να συναφεί η συμφωνία, να συμφωνήσουμε το συντομότερο δυνατό και αν δεν Υπαρκούν αυτοί οι λόγοι. Τελειώνοντα, θα πω ότι τη στιγμή κατά την οποία εμεί στις Βρυξέλλε έχουμε μείον τρει βαθμού, στη Βραζιλία έχει 30 βαθμού. Πιστεύω λοιπόν ότι όλοι θα κερδίσουμε αν μπορούμε πιο εύκολα όλοι να ταξιδεύουμε προ τη Βραζιλία. Ευχαριστώ. Thank you, Thank you. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Τικάου για το σχέδιο έκθεσης. Έχω κάποια σχόλια και ένα ερώτημα όσον αφορά την έκθεση. όπω όλοι γνωρίζουμε, μετά τη συνθήκη τη Αβώνα το Κοινοβούλιο έχει περισσότερα δικαιώματα όσον αφορά τι συμφωνίε για τι αερομεταφορέ, Η Άλτε καλωσορίζει την Συμφωνία για αερομεταφορέ Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Βραζιλία. Βραζιλίας. Θέλουμε να καταλήξουμε σε λύση που θα καλύπτουν ίδιου κανόνε από τα κράτη-μέλη και θα αντικαταστήσει τι διμερεί συμφωνίε. βασικό στόχο τη Άλτε είναι η ασφάλεια των επιβατών και των μεταφορών εν γέννη. Καλωσορίζουμε τη συμφωνία όσον αφορά τον ανταγωνισμό και που είναι υποφελής για τους επιβάτες. Υπάρχει ερώτημα που μοιάζει με τη συμφωνία τον Καναδά. Αφορά το άρθρο 4. Το Συμβούλιο έχει δικαίωμα να τροποποιεί συμφωνίες χωρίς να περνά μέσω του Κοινοβουλίου. Η νομική υπηρεσία λέει ότι αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Η κυρία Τσεκάου, μπορεί, να, κυρία Τσεκάου, μπορείτε να επεκτείνετε, να αναλύσετε περισσότερο αυτό το θέμα και να μας εξηγήσετε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια την κυρία Τσεκάου για την έκθεσή της και για τα αναλυτικά της σχόλια. Δεν θα επαναλάβω τα πάντα. Περιέγραψε πλήρως τα ωφέλη της συμφωνίας. Τρεις είναι οι γύροι των διαπραγματεύσεων. Το θέμα της διευθυνσίας και του ελέγχου το καλύψαμε και η συμφωνία για την ασφάλεια είναι καθοδόν προς ολοκλήρωση. Και συμφωνία όσον αφορά για τις τέσσερις ελευθερίες επίσης. Μπορούμε να έχουμε πρόσβαση και στη Βόρεια Αμερική, να κινηθούμε προς Βόρεια Αμερική, τώρα δεν είμαστε στη Νότια Αμερική. Ίσως εδώ να καλύψουμε και κάποια θέματα που αφορούν και τις σχέσεις με τη ΣΥΠΑ με την πάροδο του χρόνου. Έχει, υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Πρέπει να κινηθούμε γρήγορα. Εκ μέρους του ECR λέω ότι θα υποστηρίξουμε την εισηγήτρια και θέλουμε να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατόν. Η εισηγήτρια αναφέρθηκε σε όλα τα ωφέλη, τα πλεονεκτήματα. Δεν έχουμε κάτι περίπλοκο μπροστά μας. Υποστηρίζουμε τις απόψεις της. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κ. Μπουργκέλη Βενέα από Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Τσικάου για την έκθεσή της και την σύστασή της. Δηλαδή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει αυτή τη συμφωνία. Η κυρία Τσικάου σωστά υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η Βραζιλία ως οικονομικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να προσθέσω και αυτό είναι κάτι το οποίο και η κυρία Φώστερ και ο κύριος Τεσέρα το ανέφεραν. Είναι σημαντική αυτή η συμφωνία διότι είναι η αρχή μίας διαδικασίας ενίσχυσης της ε, συνεργασίας σε θέματα αερομεταφορών μεταξύ Ένωσης και ε, Βραζιλίας για ανταλλαγές ε, για την κινητικότητα των ατόμων και εμπορικού και οικονομικού ενδιαφέροντος είναι αυτή η συμφωνία. Διότι έχουμε να κάνουμε με κράτος το οποίο πληθυσμός είναι σημαντικός, όπως η Κίνα, όπως η Ιαπωνία. Έχουμε λοιπόν να προσθέσουμε ότι έχουμε πάρα πολύ, κάνει πάρα μεγάλη ε, πρόοδο το θέμα της συμφωνίας για θέματα ασφαλείας και αυτή τη στιγμή συνεχίζουμε την ε, συμφωνία με τη Βραζιλία για τις ε, υπηρεσίες αερομεταφορών. Και η μεγάλη βεβαίως εγγύηση είναι ότι οι διμερείς σχέσεις θα ευθυγραμμιστούν με το υπάρχον κοινοτικό δίκαιο. Καταλαβαίνω την παρατήρηση κυρία Σαβισάρ για το θεσμικό σκέλος του προβλήματος. Θα ήθελα όμως να ε, της πω το εξής και να πω και στην Επιτροπή σας ότι δεν μπορεί να υπάρξει αλλαγή αυτής της συμφωνίας ή οποιασδήποτε άλλης μελλοντικής συνομίας χωρίς την ε, επίσημη θεσμική παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έτσι όπως το προβλέπει η Συνθήκη της Λισαβόνας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε την κυρία Τσικάου. Σας ευχαριστώ που δώσετε το λόγο για να την ευχαριστήσω μεταξύ άλλων. Ευχαριστώ. Ίσως υπάρχει κάποια σύγχυση μεταξύ αυτής της έκθεσης και τη έκθεση για την ε, ασφάλεια. Ίσως η συνάδελφος αναφερόταν στην ε, έκθεση η οποία ασχολείται με τα θέματα ασφαλείας. Ε, πλαίσιο, ε, νομική βάση άρθρο 4. Δεν πρόκειται περί αυτού του θέματος. Κυρία Τσικάου, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά τις Διεθνείς Συμφωνίες της Αέριες Μεταφορές, μιλούμε για τρεις διαφορετικές συμφωνίες. Πρώτα απ' όλα, οριζόντια συμφωνία πλαίσιο, όπως αυτό που συζητήσαμε για τον Καναδά σήμερα το πρωί, συζητούμε μια δεύτερο είδο συμφωνίας που αφορά την ασφάλεια των πτήσεων. Αυτό είναι άλλη συμφωνία με αποκλειστική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεται να εμπλακούν τα κρατημέλη. Και τρίτου είδους συμφωνία. Αυτό, αυτή τη συμφωνία. Διότι σε ήδη υπάρχουσες διμερείς συμφωνίες που έχουν υπογράψει κράτη-μέλη και τρίτη χώρα προστίθενται βάσει κοινοτική αυτή συμφωνίας και πολλά άλλα πλέον εκτίματα. Έχουμε δηλαδή εδώ ευθυγράμμιση όλων με την κοινοτική νομοθεσία. Εναρμόνιση δηλαδή και εξασφάλιση σωστών όρων ανταγωνισμού ώστε να μην υπάρχουν διακρίσεις μεταξύ των διαφόρων ε, φορέων των κρατών μελών. άρθρο, το άρθρο 4 που αναφέρθηκε η συνάδελφος αφορά τα θέματα ασφαλείας για την ε, πολιτική αεροπορία και υπάρχει στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας ένα άρθρο το οποίο λέγει ότι οποιαδήποτε αλλαγή δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο αν υπάρχει συμφωνία των δύο εμπλεκομένων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για την παρεμβάσεις τους. Πιστεύω ότι πρόκειται για μια σημαντική συμφωνία. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό οι παρούσες διμερείς συμφωνίες να εναρμονιστούν. Γι' αυτό συνιστώ στους συναδέλφους να υποστηρίξουν αυτή τη συμφωνία συγκεκριμένη περίπτωση είναι τη Βραζιλία και τις επόμενες που θα συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τροπολογίες 8 Δεκεμβρίου, ψηφοφορία στην Επιτροπή τον Ιανουάριο, ψηφοφορία στην Ολομέλεια το Φεβρουάριο. Ξεκάθαρα όλα. Οπότε τελειώσαν οι πρωινές μας εργασίες και ξεκινάμε ξανά στις 3 με τη συμφωνία με τον Καναδά και μήνυα ακρόαση για το GNSS, την εφαρμογή. Ευχαριστώ, τα λέμε στις 3. Πώς τα